Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν επιθυμείτε και δεν σας πειράζει, να αρχίσουμε. Euh, Παρακαλώ τους συναδέλφους βουλευτές να καθίσουν για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Ως πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας προεδρεύω σήμερα και αύριο euh, η πρόεδρος κυρία Μακάβαν απουσιάζει. Ξέρετε ότι είναι στη χώρα της για το δημοψήφισμα έχει υποχρεώσεις που θα γίνει ε, τις επόμενες ημέρες και μου ζήτησε να προεδρεύσω. Αρχίζουμε λοιπόν. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Την έχετε λάβει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Διαφωνείτε. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν. Έχω μια ομάδα επισκεπτών εδώ, από τη Νέα Καλλιδονία, φοιτητέ, οι οποίοι σπουδάζουν στη Γαλλία στο Μοπελιέ. Είναι στα έδρανα των επισκεπτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω δύο ανακοινώσει πάρα πολύ θλιβερέ. Πρώτον, Ο Τζανλούκα Μπονάνο, συνάδελφός μας, βρήκε τραγικό θάνατο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου σε τροχαίο δυστύχημα στην Ιταλία. Και θα σας πρότεινα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του. Σας ευχαριστώ. Επίσης, δυστυχώς έχω να σας ανακοινώσω έναν άλλον δραματικό θάνατο, τον οποίο σίγουρα θα έχετε μάθει ήδη. Είναι η Βρετανή ε, βουλευτής Τζο Κόξ που κατέληξε την περασμένη 5η 16 Ιουνίου στα τραυματά της μετά από επίθεση που δέχτηκε στο παρελθόν ήταν βοηθός της πρώην συναδέλφου Γκλένης Κίνοκ και εργάστηκε σε θέματα της δικής μας Επιτροπής. Θα ήθελα επίση να σας προτείνω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της κυρίας Κόξ, αλλά προηγουμένως και κατ' εξαίρεση θα ζητούσα και κατόπιν αιτήματο της κυρίας Μάκαβαν, της Λίντα, που ήξερε πάρα πολύ καλά την Τζο Κόξ, να δώσω το λόγο στην ΑΝ, τμήματάρχη της Επιτροπής μας, που είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί της. Παρακαλώ, αν έχεις το λόγο. When Λοιπόν, η Τζο Κόξ εργάστηκε στην Επιτροπή μας πριν παντρευτεί, την ήξερα, ε, ως κοινοβουλευτική βοηθό της κυρίας Κίνοκ. Επειδή ήταν μέλος ε, του προσωπικού θεώρησε η Λίντα Μάκαβαν να πούμε δύο λόγια για εκείνη. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαία στη συνεργασία της, ήταν πάρα πολύ εγκάρδια, ε, πάντα χαρούμενη, ε, ήθελε πάντα να βοηθήσει, ήταν πολύ έξυπνη, απολύτως αποτελεσματική και Είχε τεράστια θαυμασική δυνατότητα και ικανότητα να εργάζεται πάρα πολύ σκληρά. Κάτι που είναι πιο σημαντικό όμως για μας είναι ότι, και ήταν προφανές προς όλους, ότι τη χαρακτήριζε ένα πάθος πραγματικά για αυτό που κάνουμε εμείς εδώ την αναπτυξιακή πολιτική. Και όταν έφυγε, και όλοι λυπηθήκαμε πάρα πολύ που έφυγε, πήγε στην Oxfam για να μπορέσει να συνεχίσει την ίδια δουλειά που έκανε εδώ της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και μόλις πριν ένα χρόνο είχε εκλεγεί στη Βουλή των Κοινοτήτων, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, εκεί ε, εξακολούθησε να εργάζεται στον ίδιο τομέα. Δεν ήταν προφανώς το μόνο που έκανε, γιατί ήταν πάρα πολύ δραστήρια σε πολλούς τομείς, αλλά κέρδισε τη φήμη της από την υποστήριξη των ε, σύρων προσφύγων, που είναι επίσης κάτι άλλο ε, με το οποίο ασχολείται ενεργά η δική μας Επιτροπή. Ε, αυτό ήταν μια παράφορη βία ε, και μια πράξη τελείως αδικαιολόγητη που έκοψε το νήμα της ζωής της και πραγματικά έστειλε κύματα τεράστιου σοκ όπου συγκλονίστηκε όχι μόνο η πολιτική κοινότητα αλλά και γενικά η κοινωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και προφανώς εντυπωσίαζε όλους εκείνους με τους οποίους συνεργαζόταν, διότι πάρα πολύ, πάρα πολύ, είπαν πάρα πολλά, πολύ αξιόλογα για την ίδια τι τελευταίε μέρε. Εγώ τι να προσθέσω. Ήθελα να σας πω μόνο ότι αυτό που έχασε τούτη η Επιτροπή είναι κάποιον που συμμεριζόταν τα οράματά μας και την αγωνία μας για την καταπολέμηση της φτώχειας, ε, για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και αυτό τα κάνει με απεριόριστη χαλήνοτη ενέργεια. Και όχι μόνο αυτό, χάσαμε και μια παλιά φίλη. Κύριος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αν. Σας προτείνω λοιπόν να τηρήσουμε ενός λεπτού και στη μνημή της Τζοκόξ. Merci. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο 3 στην ημέρηση. Η διάταξη είναι στον πρακτικό των συνεδριάσεων. Έχετε λάβει τα πρακτικά των συνεδριάσεων 9 και 10 Νοεμβρίου 2015, καθώς επίσης και τις 20 και 21 Απριλίου. Αν έχετε σχόλια για τα πρακτικά αυτά, παρακαλείστε να τα δηλώσετε στη γραμματεία μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Διαφορετικά θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά ως έχουν. Σημείο 4. Έγκριση αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών. 24 Μαΐου 2016. Και πάλι έχετε λάβει συστάσεις και αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές 24 Μάιο. Αν έχετε σχόλια σχετικά, παρακαλείστε να το υποδείξετε τη γραμματεία μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Διαφορετικά θα εγκριθούν όσοι έχουν αυτά οι αποφάσεις και οι συστάσεις των συντονιστών. Σημείο 5. Ανακοινώσεις Επιτροπής. Δεν ξέρω αν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχόλια, ανακοινώσει, δηλώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια μικρή υπενθύμηση για ε, δύο μεγάλες ανακοινώσεις στις οποίες ε, ε, ενέχεται η δική μας Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ ενέκρινε το νέο πλαίσιο στις 6 Ιουνίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία με τις χώρες και για τη μετανάστευση και στις 8 του μηνός ενέκρινε τη στρατηγική για ε, διεθνείς πολιτιστικές θέσεις. Και αυτά τα δύο έχουν, θέση, έχουν και σχέση με τη δική σας Επιτροπή και τη δική μας Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Σημείο 6 της τη διάταξης. Λάβαμε μια ερώτηση από τον συνάδελφο Ερίκε Γκερέρο Σαλόμ για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες ε, για την Τουρκία. Το θέμα αυτό είναι γεγραμμένο στην ημερήσια διάταξή μας. Και θα δώσω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση. Νιέρ και Έκο. Ε, έχω. Δεν ξέρω ποιο θέλει πρώτο το λόγο. Έκο, ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά και ο συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Νιέρ θα συμπληρώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρα Σαλόμ για την ερώτηση αυτή, η οποία μα δίνει τη δυνατότητα μέσα σε λίγα λεπτά να ενημερώσουμε στο δυνατόν πληρέστερα την Επιτροπή σα για την υλοποίηση αυτή τη διευκόλυνση αυτού του μηχανισμού. Δεν χρειάζεται να σας πω τα γενικά. Αυτός ο μηχανισμός εντάσσεται στη Γενική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και όπως λέει και το όνομα διευκόλυνση, υποτίθεται ότι διευκολύνει ε, τα συμπεφωνημένα. Δηλαδή ε, συντονισμός ε, ορισμένων προϋπαρχόντων μέτρων και μηχανισμών που είχαν να κάνουν ορισμένα με την ανθρωπιστική βοήθεια και άλλα με την πολιτική γειτονία. Και αυτό εξηγεί την πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων. Επίσης πρόκειται για ένα μέσο συντονισμού μεταξύ οικονομικών ε, συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αφενός και από τα κράτη-μέλη αφετέρου. Οι οικονομικές συνεισφορές από τα κράτη-μέλη πηγαίνουν στον ε, κοινοτικό προπολογισμό με βάση μια προκαθορισμένη κλίδα που είχε αποφασίσει το Συμβούλιο και μπορούμε να σας ενημερώσουμε ότι επί του παρόντος το σύνολο αυτών ε, των συνεισφορών, των εισφορών αυτών έχουν ε, καταβληθεί το συνολικό ποσό που προβλέπεται για αυτή τη διευκόλυνση για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο μπορεί και να διπλασιαστεί για τα επόμενα δύο οικονομικά έτη, άρα από 3 να είναι 6 δις το ποσό αυτό, εφόσον βέβαια οι όροι της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ε, τηρηθούν και εφαρμοστούν πλήρως. Η υλοποίηση αυτού του μηχανισμού διευκόλυνσης ε, γίνεται αντικείμενο συντονισμού από μια επιτροπή διοικούσα επιτροπή, steering committee μπορούμε να την πούμε, ε, που απατήσει τα εκπροσώπηση των κρατών μελών. Η Τουρκία εκπροσωπείται επίσης ως παρατηρήτρια χώρα όμως. Και η Επιτροπή αυτή δεν είναι ε, διαχειριστική επιτροπή, αλλά συνοδευτική θα την χαρακτήριζα. Είναι ένα είδος πλατφόρμας όπου οι γενικές κατευθύνσεις που αφορούν την εφαρμογή του μηχανισμού διευκόλυνσης ε, που βάλλονται στα κράτη-μέλη, σημαντικούς ε, συνεισφέροντες στην υλοποίηση αυτού του μηχανισμού υπογραμμίζω και συχνά γίνονται αναφορές ότι αφορά την υλοποίηση αυτού του μηχανισμού ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν ενδεχομένως να ασκήσουν ε, ρόλο επιτήρησης, παρακολούθησης και να επιβάλλουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιους όρους. Η κατανομή των συνολικών ποσών μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής γειτονίας είναι ενδεικτική. Ένα δις επί των τριών, το ένα τρίτο δηλαδή του ποσού του συνολικού προορίζεται για την α, αμυγός ανθρωπιστική βοήθεια και τα άλλα δύο τρίτα, τα δύο δις δηλαδή, προορίζονται για την υλοποίηση μέσω αναστοπλές τη πολιτική ε, ανάπτυξη και γειτονία. Είναι ένα ποσό ενδεικτικό όμω παραλαμβάνω. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να τονίσω και κάτι ακόμη. Αυτά τα κονδύλια διατίθενται με βάση τους κανόνες και σύμφωνα με την νομική βάση του χρονομοτοδοτικού μέσου. Η Συνοδευτική Επιτροπή, αυτό το Steering Committee, είναι Συνοδευτική Επιτροπή, δεν αποφασίζει, είναι μια Επιτροπή υποστήριξης όταν θα έχουν συμφωνηθεί οι στρατηγικές, γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις από αυτήν την steering committee έπειτα η Κομισιόν είναι αυτή η οποία θα πρέπει να εφαρμόσει αυτές τις γενικές κατευθύνσεις στην πράξη με τους νομικούς διάβλους, ε, τους πλέον κατάλληλους και την ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλουμε τα κονδύλια να χορηγούνται αυστηρά με βάση τον εφαρμοστέο για την ανθρωπιστική βοήθεια χρηματοδοτικό κανονισμό. Το ίδιο θα ισχύσει αύριο για την πολιτική γειτονία και ούτω καθεξής. Η Επιτροπή αυτή τώρα, ε, υποστήριξη, steering committee, έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές και θα συνεδριάσει για τρίτη φορά στα τέλη του μήνα. Και να σας πω ότι στις δύο πρώτες της συνεδριάσεις ενέκρινε ένα στρατηγικό έγγραφο που είχαν προτείνει οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο βασίστηκε στην αξιολόγηση των αναγκών ε, needs assessment που έγινε σε βάθος και σε στενή συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Το εν λόγω στρατηγικό έγγραφο εντοπίζει έξι προτεραιότητες. Ανθρωπιστική βοήθεια, αμυγεγός, εκπαίδευση, διαχείριση μεταναστευτικών ροών, υγεία, υποδομές σε τοπικό επίπεδο και στήριξη της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Και όλα αυτά εφαρμόζονται με πρωτοβουλίες και με προγραμματικά έγγραφα αφήνω τώρα το λόγο στο συνάδελφό μου, ο οποίος θα σας ενημερώσει πιο συγκεκριμένα για τις προτεραιότητες ε, της πολιτικής γειτονίας. Κατανοώ ότι η ερώτηση του κ. Γκερέρο Σαλόμ βέβαια εστίαζε κυρίως σε ό,τι άπτεται της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δηλαδή στο ανθρωπιστικό σκέλος του μηχανισμού διευκόλυνσης. Το συνολικό ποσό δεν θα σας διέφυγε ότι δημοσιεύθηκε προσφάτως ε, το έγγραφο Humanitarian Implementation Plan, HIP, για την Τουρκία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις αρχές του Ιουνίου δημοσιεύθηκε το έγγραφο αυτό και αν το διαβάσετε θα βρείτε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τις γενικές αυτές κατευθύνσεις που σας περιέγραψα. Η ανθρωπιστική βοήθεια για το τρέχον οικονομικό έτος θα βασιστεί σε τέσσερις διαφορετικές προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα, και νομίζω ότι ήταν και η ανησυχία και του κύριου, του κύριου Γκερέρο Σαλόμ, ο στόχος μας, αν μου επιτρέπετε τον όρο, τέλο πάντων είναι τόσο δόκιμο, σας πω η προτεραιότητά μας είναι η πρόσφυγες που δεν φιλοξενούνται σε κάποιο καταβλισμό. 10% περίπου μόνο των προσφύγων που έχουν καταγραφεί σε τουρκικό έδαφος φιλοξενούνται σε καταβλισμούς προσφύγων. Οι υπόλοιποι είναι διάσπαρτοι ε, στην όλη περιοχή, κυρίως εκεί γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Για αυτούς κυρίως, για αυτόν τον πληθυσμό ε, σε αυτόν έχουμε εστιάσει κυρίως. Και σίγουρα εφαρμόσουμε τις βασικές αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας, άρα θα εστιάσουμε και στις πλέον ευάλωτες ομάδες μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Τι κάναμε μέχρι τώρα. Επεκτείναμε και διευρύναμε κάποια προγράμματα ήδη ισχύοντα ε, για την κάλυψη βασικών αναγκών ε, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και συγκεκριμένα διανομή τροφίμων, στέγαση, μέτρα υγιεινής κτλ. Αυτή ήταν η πρώτη μας ε, συνεισφορά που ε, καλύπτεται από συμβάσεις της τάξης ε, των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, η δεύτερη φάση που έχει ξεκινήσει είναι ένα πολύ φιλόδοξο σύστημα διανομής ε, χρήματος, ε, ρευστού χρήματος που θα ξεκινήσει. Εστιάζουμε πάλι εδώ στις πλέον ομάδες, στον πληθυσμό στόχο εντός εισαγωγικών, που θα είναι περίπου ένα εκατομμύριο δικαιούχοι αυτοί για το οικονομικό έτος 2016-2017. Τρίτη προτεραιότητα, συμπληρωματική με την προηγούμενη, είναι ορισμένε δραστηριότητες ε, σε ό,τι αφορά την προστασία των προσφύγων, συμπληρωματικά προσώπη ό,τι κάνουν οι συναδελφοί από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ γειτονία, εκπαίδευση ε, σε συνθήκες έκτακτης ε, ανάγκης, education in emergency. Αυτό είναι προτεραιότητα του Επιτρόπου στη Λιάννη, όπω γνωρίζετε και ήδη σας παρουσίασε τα σχετικά, απαντώντα και στις ερωτήσεις σας. Το ίδιο Ισχύει και για την παρέμβασή μας στην Τουρκία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι η προστασία κατά της βίας σε βάρος γυναικών, προστασία σε ομάδες ευάλωτες, σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπήρεια κτλ. Ε, Φιστώ επίσης την προσοχή σας στο ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα απευθύνεται σε όλους τους καταγεγραμμένους πρόσφυγες, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Δεν περιορίζεται σε Σύρους μόνο πρόσφυγες. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε και πρέπει να το είχα πει από την αρχή ίσως. Τελευταία προτεραιότητα, μόλις ε, σας προείπα ότι η δική μας ε, παρέμβαση αφορά κυρίως αυτούς που δεν φιλοξενούνται σε κάποιο ε, καταβλισμό προσφύγων, αλλά και στους καταβλισμούς πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, γιατί οι πρώτοι καταβλισμοί έγιναν σε ένα πολύ πρώιμο ε, αρχικό στάδιο της κρίσης. Προοδευτικά λοιπόν οι εγκαταστάσεις ε, χαρακτηρίστηκαν από κόποση, θα μπορούσα να πω, και έχουν απαρχαιωθεί πλέον. Εμείς θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε θεωρηθεί από προτεραιότητα σε σχέση με άλλε μα προτεραιότητε. Όμω, εξετάζουμε και αυτό το ενδεχόμενο, να αυξήσουμε δηλαδή την υποστήριξή μα προ τι υπηρεσίε που παρέχονται στου πρόσφυγε σε καταβλισμού πρόσφυγων, ώστε και οι τουρκικέ αρχέ να μπορέσουν να αφιερώσουν τα απαιτούμενα ποσά για την ε, ανακαίνιση και τον εξυγχρονισμό αυτών των καταβλισμών. Αυτή είναι μια πρώτη σειρά απαντήσεων, κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθω φυσικά εφόσον ο κύριος Γκερέρο Σαλόμι, άλλοι βουλευτές επιτροπή σας έχουν απορίες ή θέλουν πληροφορίες. Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου που εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση για την Πολιτική Γειτονία. Σε ευχαριστώ. Thank you very um, um, ευχαριστώ πολύ κύριος Ζεμπρό ήταν πολύ ε, περίεκτικός. Εγώ απλά θα σας δώσω μία εικόνα ε, όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτής της διευκόλυνσης. Είναι τμήμα της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του Μαρτίου ε, είναι πλήρως λειτουργική, έχουμε λάβει συμβολές από όλα τα κρατημέλη και έχουμε καταχωρήσει μέχρι στιγμής 750 εκατομμύρια. Έχουμε κάνει συμβάσει 150 και έχουμε διαθέσει 105 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρώσουμε υπό το τμήμα το αναπτυξιακό αυτής της διευκόλυνσης ένα ειδικό μέσο, ένα πακέτο μέτρων που θα βοηθήσει τους πρόσφυγες στην Τουρκία, εστιάζοντας την παιδεία, την υγεία, τη δημοτικές υποδομές και την κοινωνική και οικονομική βοήθεια συμπληρώνοντας ε, κάποια πρώιμα ειδικά μέτρα που είχαμε υιοθετήσει τον Απρίλιο για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες που επιστράφηκαν στην Τουρκία για να τους δώσουμε στέγαση ε, υγειονομική περίθαλψη και τρόφιμα. Και επίσης για να συμπληρώσουμε ένα προηγούμενο μέτρο ώστε να ενισχύσουμε τις ε, δυνατότητες της τουρκικής ακτοφυλακής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής, ιδιαίτερα τον κύριο Ντεμπρού, για τις ε, πολυάρσεις πληροφορίες που μας έδωσε σε σχέση με την ερώτηση που εγώ έθεσα. Θα πρέπει να τονίσω ότι, όπως γνωρίζετε κι εσείς άλλωστε, ότι εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν Είμαστε σχετικά επικριτικοί και σε ορισμένε περιπτώσει και πολύ επικριτικοί απέναντι σε αυτή τη συμφωνία που επετέφθη με την Τουρκία. Ωστόσο, αυτό που θέλουμε εδώ δεν είναι το να συζητήσουμε αν είναι κατάλληλη ή όχι αυτή η συμφωνία, αλλά να παρακολουθήσουμε από την προοπτική του Κοινοβουλίου την, το κατά πόσο εφαρμόζεται ή όχι. Και από αυτή την άποψη έχετε να μας φέρετε μάλλον καλά νέα Δηλαδή, προστατεύεται οποιοδήποτε είναι σε αυτή την κατάσταση πρόσφυγα και που το έχει αυτό ανάγκη, είτε είναι Σύριος είτε όχι. Δηλαδή έχουμε και στόχο προτεραιότητας όλες τους ευάλωτους πληθυσμούς και έχουμε και ένα συγκεκριμένο τμήμα που απευθύνεται στις, στις επίγουσες καταστάσεις. Όλα αυτά είναι, θέματα, είναι θέσεις μάλλον που εγκρίθηκαν σε διάφορες συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα ήθελα μόνο να θέσω μια επιπλέον ερώτηση, δηλαδή μέχρι ποιου σημείο οι τουρκικές αρχές συνεργάζονται με την εφαρμογή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη συμφωνία και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτούς τους πληθυσμούς που δεν είναι συγκεντρωμένοι σε καταβλισμούς, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αλλά είναι σκόρπιες ανάμεσα στον πληθυσμό. Δεδομένου ότι στο καταστατικό των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις Τουρκίες, μάλλον το καθεστώς των ε, ΜΚΟ στην Τουρκία είναι κάπως ασαφές <laughs> και μπορεί να ε, καταστήσει αυθαίρετη την απόφαση πρόσβασης προς αυτούς τους πυρήνες, τους θύλακες μάλλον ε, πληθυσμού. Ευχαριστώ λοιπόν για τις πληροφορίες. Δεύτερον, έχουμε κοινέ προτεραιότητες και τρίτον, ε, θέλω να διευκρινίσω όσον αφορά τη συμπεριφορά των τουρκικών αρχών, όσον αφορά τη διευκόλυνση πρόσβασης ε, για τις ΣΜΚΙΟ, που ασχολούνται με την εφαρμογή αυτής της ίδιας συμφωνίας, πρόσβασης στους πληθυσμούς, στους θύλακες που το χρειάζονται. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Θέλετε να απαντήσετε πολύ σύντομα, σας παρακαλώ, πολύ σύντομα. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο και ευχαριστώ τον κύριο Γκερέρο Σαλόμ για την θετική του αξιολόγηση. Το είπα και πριν από λίγο, εργαζόμαστε ότι η κυβέρνηση και οι τουρκικές αρχές έχουν συμβουλευτικό καθεστώς όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της διευκόλυνσης με την εξαίρεση των όσων αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί ήμασταν σαφείς απέναντι στους συνομιλητές μας, τους το είπαμε η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αυτό που είναι. Δηλαδή περνά μέσα από μη κυβερνητικού ε, φορείς, ε, ΟΗΕ, ΜΚΟ, ε, Ερυθρό Σταυρό Διεθνή Επιτροπή και Ερυθρή Μισελίνος που είναι πολύ επαγγελματικοί και αποτελεσματική οργάνωση και γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα κριτήρια της, ε, του πόσο ευάλωτοι είναι κάθε φορά οι πληθυσμοί. Έχουμε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Για παράδειγμα, το σύστημα ε, εμβασμάτων ε, με διάφορους σκοπούς είναι ένα σύστημα το οποίο το επεξεργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με το τουρκικό Υπουργείο γιατί στόχο έχει από τη στιγμή που θα φτάσει η διευκόλυνση στην Τουρκία να ενταχθεί στο σύστημα το τουρκικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη διάρκεια του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής καταγράψει προβλήματα πρόσβασης. Είχαμε προβλήματα άλλου είδους, αλλά όχι, δεν ήταν αυτή η ερώτηση του κ. Γκέρερος, όσον αφορά ε, υποθέσεις στα σύνορα και από τη μια και από την άλλη πλευρά των συνόρων με τη Συρία. Και είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να καταστήσουμε σαφές στους Τούρκους συνομιλητές μας και μέχρι στιγμής ο διάλογος λειτουργεί και οι συμβάσεις για τις οποίες σας μιλούσα για όσον μας αφορά εμάς έχουμε ήδη κάνει συμβάσεις 160 εκατομμύρια ε, ευρώ ε, με συμβάσεις ε, με διάφορους εταίρους μεταξύ των οποίων και ΜΚΟ που έγιναν δεκτές που μάλλον γνωστοποιήθηκαν προς τις τουρκικές αρχές. Δεν χρειάζονταν έγκριση από πλευράς τουρκικών αργών. Αυτά, Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ και θα σας πρότεινα να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη του υπαριθμών 7 φόροι κατά την εξαγωγή και άλλοι περιορισμοί στις πρώτες και ο περιορισμός τους μέσω των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Ο αντίκτυπος στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για μία μελέτη. Είναι το πρώτο ουσιαστικό θέμα σήμερα. Είναι η παρουσίαση μελέτης. Μια μελέτη που αναθέσαμε για το πώς χρησιμοποιούνται οι φόροι σε εξαγωγές και άλλε επιστροφέ σε πρώτε ύλες και πώς περιορίζονται από τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και πώς επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε τον κύριο Σάμουελ Σούμπερτ από το Πανεπιστήμιο Webster, Webster στη Βιέννη, ε, που είναι ένας από τους συντάκτες αυτής της μελέτης. Θα μας παρουσιάσει τα πορίσματα και τις συστάσεις του δίνω αμέσω το λόγο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Παρακαλώ κύριε Σούμπερτ, έχετε το λόγο. Merci beaucoup, Monsieur Ευχαριστώ πολύ κύριε Πονγκά. Κυρίε και κύριοι, μέλη τη Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή, σας ευχαριστώ πολύ. Sorry to switch to what is a, rather theoretical... Ε, αυτό μπορεί να είναι θεωρητικό ζήτημα και ανιαρό σε σχέση με αυτά που αναφέραμε προηγουμένω, που ήταν για μένα συναρπαστικό. οι φοιτητέ ε, στα πίσω έδρα να θα γνωρίζουν αυτά που πρόκειται να σας πω εγώ να καλύψω ε, και που ήταν αντικείμενο της μελέτης μας. Με δύο λόγια, τι κοιτάξαμε, τι μελετήσαμε, κατά πόσο και σε ποιο βαθμό οι φόροι και οι περιορισμοί στις εξαγωγές είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και αν ναι, θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη και την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό είναι το αντικείμενο και το πρίσμα από το οποίο το κοιτάξαμε. Μπορεί κανείς να το δει από την οικονομική σκοπιά, αλλά εκτός αυτού έρχεται να προσθεθεί και ένα άλλο στοιχείο που είναι η αναπτυξιακή πτυχή. Γιατί έχω πολλά χρόνια δραστηριότητα σε αυτό το τομέα και στην εφαρμογή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πάμε λοιπόν, αν θέλετε, στην πρώτη διαφάνεια. αυτή ακριβώς. Λοιπόν, με δύο λόγια. Θα τα γνωρίζετε πολλά από αυτά που θα ακούσετε ενδεχομένω. Γνωρίζουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρησιμοποιούν τους φόρους στην εξαγωγή προϊόντων και τους περιορισμούς διαφόρων ειδών για διάφορους τρόπους. Μεταξύ αυτών είναι να σταθεροποιηθούν οι τιμές εγχώριες, να αναπτυχθεί η βιομηχανία η προστιθέμενη αξία δηλαδή στο εσωτερικό της οικονομίας τους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πολύ συχνά σημειώνουν οι χώρες αυτές είναι να αποκτήσουν εισόδημα ε, ε, ως πόρους κρατικούς. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί. Και το άλλο είναι διτό. Από τη μια θέλουν να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό, αλλά από την άλλη να ε, εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν την αηφορία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Και συνήθως αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Εκείνοι που ζητούν λοιπόν να επιβάλλονται φόροι κατά την εξαγωγή των ε, προϊόντων έχουν λόγους πάρα πολύ εύλογους να το επιθυμούν να το ισχυρίζονται. Πρώτον, αυτά είναι εύκολα χρήματα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, αν βάλεις ένα χώρο στην εξαγωγή προϊόντων, ε, είναι πολύ καλός τρόπος να μαζεύει λεφτά η κυβέρνηση, ιδιαίτερα όταν είναι εύκολη η συλλογή τους. Για λόγους που θα εξηγήσω στη συνέχεια, πολύ συχνά ε, συνδέεται με πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα. Μπορεί να μην είναι η σταθερότητα που εσείς επιζητείτε, δηλαδή με την έννοια της αναδιανομής, αλλά δεν είναι το χάος. Και το κλασικό είναι προστασία από ε, ανταγωνισμό από άλλες ε, εταιρείες. Στην αρχή όταν ε, ξεκινήσαμε τέθη το μεγάλο ερώτημα. Όλα αυτά είναι άραγε νόμιμα. Και τι λέει η πραγματικότητα. Στο διεθνές εμπόριο οι κανόνες δεν απαγορεύουν την επιβολή φόρων στην εξαγωγή. Βέβαια, για να μην, να μην σταματάνε και τελείω τι εξαγωγέ, να μην είναι τόσο υπερβολικές ώστε να παραλύει. Και υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί στις εξαγωγές ε, και κανόνε, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλέ εξαιρέσει για του κανόνε αυτού. Τι βλέπουμε λοιπόν. Όταν κανείς περιορίζει τη δυνατότητα μιας χώρας να επιβάλλει φόρους ή περιορισμούς στην εξαγωγή, πρέπει να κοιτάξουμε ότι μπορεί αυτό να έχει και αρνητικές επιδράσεις στις χώρες αυτές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους στόχους τους αναπτυξιακούς. Εγώ τι έκανα λοιπόν, έχω οργανώσει τις επόμενες διαφάνειες ε, και τις έχω εντάξει σε αυτούς τους ε, τομείς, έσοδα για την κυβέρνηση, αναπτυξιακή ε, βοήθεια, σταθεροποίηση των τιμών, περιβάλλον κτλ. Και πρώτα συγκρίνω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τι κάνει το διεθνές στερέωμα. Και ποια είναι η αποτελεσματικότητα όλων αυτών. Και το τι θα συνέβαινε από πρακτική σκοπιά αν γίνουν πιο σφιχτοί οι κανόνες και αρθούν οι φόροι αυτοί. να δούμε ενδεχομένως κάποιες εναλλακτικές λύσεις και συστάσεις. Προσπάθησα να το κάνω όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Ξέρω, μερικοί από εσά θέλετε περισσότερους περιορισμούς και άλλοι να καταργηθούν τελείως. Κάπου στη μέση θα βρεθώ εγώ. Στα αγγλικά υπάρχει μια παροιμία που λέει ε, ότι δεν έχω σκύλο σε αυτή τη σκυλομαχία, δηλαδή ότι δεν έχω ιδιαίτερο συμφέρον ε, ούτε ε, έχω ιδιαίτερη θέση, δεν έχω σκύλο σε αυτή την κοινομαχία. Ε, δεν, δεν έχω ιδιωτελή ξέρω κριτήρια ή σκοπούς. Απλώς το εξετάζουμε από τις δύο σκοπιές για να κάνουμε τη συζήτηση και να δούμε πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν λοιπόν διεθνείς συμφωνίες ΓΑΤ, POE, που καταρχήν απαγορεύουν ε, τους ποιοτικούς, ποσοτικούς μάλλον περιορισμούς, αλλά επιτρέπουν κάποιες ε, εξαιρέσεις σε ειδικέ περιστάσεις. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιους ελέγχους ε, νομίσματος. Από την άλλη, οι φόροι κατά την εξαγωγή επιτρέπονται, δεν απαγορεύονται οι φόροι, εκτός αν είναι τόσο παράλογοι και φορομπηχτικοί που παραλύουν την εξαγωγή ενός προϊόντος. στα EPA, στις συμφωνίες αυτές της εμπορικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ισχύουν οι περιορισμοί του ΓΚΑΤ και του ΠΟΕ με κάποιες άλλες εξαιρέσεις. Στην κάρι φόρμ απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή εξωτερικών φόρων στην εξαγωγή. Με τη Δυτική Αφρική απαγορεύονται οι νέοι φόροι με κάποιες εξαιρέσεις προσωρινές. και επίσης απαγορεύεται να αυξηθούν οι συντελεστές των υπαρχόντων φόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ, απαγορεύονται οι νέοι ε, φόροι κατά την εξαγωγή, αλλά επιτρέπονται οι προσωρινές εξαιρέσεις, ε, αντίστοιχα με τα όσα ισχύουν για άλλες συμφωνίες. Και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης, SADC, νέοι φόροι απαγορεύονται με κάποιες εξαιρέσεις. Γενικά ισχύουν τα όσα ισχύουν στον ΠΟΕ. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε λίγο τι γίνεται με το σκεπτικό και το συλλογισμό. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο δικαιολογίε, αλλά αιτιολόγηση. Για ποιο λόγο επιβάλλονται, για ποιου λόγου αυτοί οι φόροι, για ποιο λόγο δεν θέλει κάποια χώρα να επιβάλλει φόρο στην εξαγωγή ενό προϊόντος. το ονόμασα η βάση για τους φόρους κατά την εξαγωγή, η λογική δηλαδή, ότι είναι η καλή πολιτική και έχει και ένα στοιχείο επιδότησης, δηλαδή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τα σύμβολα. Εύκολα τα διαβάζετε. Περί τίνος πρόκειται. Όταν αυξάνονται οι τιμές, το δέλτα είναι τιμές, ε, μειώνεται ε, το εισόδημα που έχει ο πληθυσμός και η αγοραστική δύναμη και επειδή αυτό είναι λόγος επιβίωσης, άμα τους μειώσει το εισόδημα υπάρχει πολιτική αστάθεια. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να ε, εκτοξευθούν οι τιμές και οι φόροι στην εξαγωγή κρατούν τις τιμές κάπως συγκρατημένες και υπάρχει κυκλοφορία του προϊόντος ε, και στην εγχώρια αγορά. Δεν φεύγει όλο. Ε, όταν αυξάνονται οι φόροι στην εξαγωγή, μειώνονται οι τιμές, άρα είναι προς όφελος των εγχώριων καταναλωτών και είναι πάρα πολύ δημοφιλής αυτή η φόρη. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, αν ξέρετε πώς έχει η κατάσταση με την αναπτυξιακή βοήθεια και τις οικονομίες των χωρών αυτών. Αν ξέρετε τη διατίμηση στο ψωμί και στο καύσιμο, σε ορισμένες χώρες ε, γιατί επιδοτούνται, είναι ε, τεχνητά σε χαμηλό επίπεδο γιατί αν τις άφηναν να φτάσουν σε ισορροπία ε, της αγοράς ο κόσμος θα εξεγυρώταν γιατί δεν θα είχε λεφτά να πάρει ούτε ψωμί ούτε κάψιμο. Οπότε, αυτοί οι πιο αυστηροί κανόνες τι επιπτώσεις έχουν. Ας πούμε ότι προσπαθούμε να απαγορεύσουμε ε, τους φόρους κατά την εξαγωγή να τους μειώσουμε δραστικά. Από πλευράς εγχωρίων τιμών τι θα γίνει. Είναι πολύ εύκολο με τα εμπειρικά στοιχεία που έχουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Βράχει πρόθεσμα, υπάρχει επίπτωση και σε μεγάλο βαθμό αρνητική. Αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η επίπτωση ούτε μέσο πρόθεσμη ούτε μακροπρόθεσμη. Υπάρχουν πολλές μελέτες που τα μελετούν αυτά τα πράγματα πριν αλλάξει πολιτική και μετά. Αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία με τις εγχώριες τιμές είναι το εξής. Όταν ε, καταργούνται οι εξαγωγικοί φόροι, μειώνεται το κίνητρο για να ε, παραχθεί τη θέμενη αξία. Δηλαδή, τι γίνεται. Αν δεν έχω το φόρο ε, στην εξαγωγή και δεν θέλω να κρατήσω στη χώρα την παραγωγή, πηγαίνω και εξάγω το προϊόν. Έχω μεγαλύτερο κίνητρο για να το εξάγω παρά να το κρατήσω στη χώρα. Αυτό έχει αρνητική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό όμως της οικονομίας της αναπτυσσόμενης χώρας. Και πάλι βραχυπρόθεσμα ισχύει αυτό. Για μακροπρόθεσμα δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι στην περίπτωση των τροφίμων, so, ε, στα γεωργικά προϊόντα, η μείωση της εσωτερικής προσφοράς, επειδή εξάγεται το, το προϊόν γιατί δεν έχει φόρο, αυτό θα μπορούσε να πλήξει τους πιο ασθενείς και εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Παραδείγματα έχουμε σε αυτή την περίπτωση στην Ινδονησία και την Ταϊλάνδη. Υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες ε, με φινικέλαιο και σπόρους με αποτελέσματα ανάμεικτα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι Ουκρανία, Ρωσία και το ψωμί. Τι συνέβη εκεί λοιπόν. Ήταν στη διατίμηση το ψωμί για να συγκρατηθούν οι τιμές προς τα κάτω και ήταν και σιτοβολώνες οι χώρες αυτές. Και επειδή ξαφνικά κράτησαν όλες τις ποσότητες στο εσωτερικό για να μην ανισχύει ο κόσμος, έχασαν τη θέση του στη διεθνή αγορά και ο κόσμος διεθνώς σταμάτησε να αγοράζει ψωμί βυσιτάρι ας πούμε από τη Ρωσία και την Ουκρανία γιατί δεν ήταν αξιόπιστοι προμηθευτές και αυτό είχε πολύ ανητικές επιπτώσεις και σχεδόν διαρθρωτικές, πολύ βαριές. Υπάρχουν εναλλακτικέ σε όλα αυτά τα μέτρα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Κάτι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάς για τις αναπτυσσόμενες χώρες και το εμπόριο, λες και είναι δύο πράγματα τελείως ξεχωριστά μεταξύ τους. Γιατί υπάρχουν και προγράμματα που τα συνδέουν. Okay. So, of course... Λοιπόν, ε, ε, τι θα πρότεινα. Να κοιτάξετε να υπάρχει μεγαλύτερη τεχνική συνεργασία ε, που αυξάνει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό και είναι πιο εύκολο να κρίνει κανείς την αγορά και να δημιουργηθούν συστήματα ασφάλειας, εξασφάλισης και προστασίας. Για συστήματα ασφάλειας, αποζημίωσης, δηλαδή από καιρικέ συνθήκες αντίξωες ε, ή προστασία ευρύτερη ε, ε, με τρόπο χρήματα δηλαδή ένα σύστημα futures παραγόγων που μπορεί ακόμα να μην υπάρχει στη χώρα if we go on to the next slide. Προχωρούμε στο επόμενο. Η βιομηχανική ανάπτυξη είναι αντίστοιχα τα προβλήματα. Βασικά εδώ τι έχουμε. Οι φόροι κατά την εξαγωγή βοηθάνε την προστιθέμενη αξία γιατί ακριβώς έχουν ένα στοιχείο επιδότησης. Και το πιο σημαντικό είναι και πάλι το εξής. Όταν έρονται αυτοί οι κανόνες, ο αντίκτυπος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Δηλαδή, αν καταργηθεί ο φόρος κατά την εξαγωγή, δεν σημαίνει απολύτως ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Για να λυθεί το ζήτημα της προστιθέμενης αξίας, αυτό που χρειάζεστε είναι ειδικευμένους εργάτες. Αυτό γίνεται με την κλασική ανάπτυξη, με προγράμματα μπορεί να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία και ό,τι άλλο θέλετε, αλλά τελικά δεν έρχεται από εκεί η ανάπτυξη. Χρειάζεται εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Το πιο κοινό που σας είπα ήταν ε, για, για έσοδα για το κράτος, για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυξάνεται το κρατικό εισόδημα με μικρό κόστος και χώρες που έχουν τέτοιους εξαγωγικούς φόρους και έχουν ως πηγή εισοδήματο αυτό το φόρο, δεν μπορούν να μαζέψουν τους φόρους διαφορετικά. Δηλαδή είναι κατακαιρματισμένη η οικονομία, αλλά δεν υπάρχει καλή φορολογική αρχή η ίσπραξη των φόρων και αυτός ο φόρος μπορεί να είναι η μοναδική πηγή εισοδήματο για το κράτος. Άρα το να καταργηθεί θα είχε αντίκτυπο ενδεχομένως και ολέθριο για τη χώρα. Και το καλύτερο παράδειγμα που βρήκαμε ήταν η Γουινέα που έχει αποθέματα, κοιτάσματα βοξίτη και ε, διατηρείται ο φόρος εκεί. Βεβαίως όταν έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισαγωγέ υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και ο σκοπός είναι να ε, επενδύσει κανείς σε καλύτερους μηχανισμούς διακυβέρνησης και πάντα μιλώ για την άμεση βοήθεια. Και το σημαντικότερο και το πιο δύσκολο τελικά είναι το θέμα του περιβάλλοντος. The, has been one... Το περιβαλλοντικό ζήτημα στη βιβλιογραφία αντιμετωπίζεται υπό δύο πτυχές. Το πρώτο είναι να διατηρήσουμε τους φυσικούς πόρους που υπάρχουν τα κοιτάσματα κτλ. Και το δεύτερο, να αντιμετωπίσουμε τη διάβρωση του εδάφους από την ε, υπερβολική δραστηριότητα, την κτηνοτροφική, τη γεωργική κτλ. Τι γίνεται όταν έρονται οι φόροι κατά των ε, εξαγωγών. Βλέπουμε δύο τελείως διαφορετικές μεταξύ τους ε, εκβάσεις που εξαρτώνται από το κατά πόσον η εγχώρια ζήτηση για τον λόγο προϊόν αυξάνεται ή όχι. Δηλαδή η επιτυχία ή η αποτυχία έχει ως προϋπόθεση κάτι που δεν μπορούμε εκ των προτέρων να ελέγξουμε. Το πρώτο σενάριο είναι ένα είδος ε, επιδημίας επικεντρώνονται όλοι στο ίδιο, στην ίδια πρώτη υπερπαραγωγή και μείωση του περιβάλλοντος, αν καταργηθεί ε, ο φόρος κατά την εξαγωγή, σε μικρές χώρες και οικονομίες, αν είναι τόσο πολύ ε, μικρές, δεν θα αλλάξει η ζήτηση ουσιαστικά, οπότε θα έχουμε και πολύ μικρή επίπτωση για το περιβάλλον. Θα πρέπει να βλέπουμε λοιπόν το μέγεθος ε, της εκάστοτε οικονομίας, τον προσανατολισμό, τη διαφοροποίηση της οικονομίας και αν δεν υπάρχει συστηματοποίηση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Η Κίνα μας παρέχει το καλύτερο παράδειγμα περιβαλλοντική συλλογιστική ουσιαστικά για να συγκρατήσει τις ε, σπάνιες γέες εντός. Αυτό οδηγεί ε, σε χαμηλές ε, τιμές και στην Κίνα η υπηρεσίες αξία αξίας, δημιουργεί περισσότερη ζήτηση και παράνομη εξορρυκτική δράση με τεράστια περιβαλλοντική ζημία. Άρα τα προγράμματα συνεργασίας είναι η καλύτερη δημιουργική. για να ολοκληρώσω, All Όλες οι συστάσεις ανάλογα από το που βρίσκεται κανείς και σε σχέση με τους φόρους κατά των εξαγωγών μπορούν να υποδερεθούν σε γενικές αφενός. Ε, τώρα μπορεί κανείς να ενημερώσει τους εταίρους για τις ε, αρνητικές επιπτώσεις αυτών των φόρων ε, σε σχέση με την κατάργηση, την απαγορευσή τους. Δηλαδή αν το κάνουν αυτό μεν, αλλά ίσως και με κάποιες προϋποθέσεις αυτό θα βοηθούσε. Επίσης θα έλεγα ότι η τεχνική συνεργασία ενισχυμένη πρέπει να συμπεριληφθεί. Αν μιλάμε για μια πηγή εισοδήματος, πραγματικά χρειάζεται εναλλακτική λύση, αλλιώς η κυβέρνηση θα πέσει σε ελεύθερη πτώση. Υπάρχει μια διαφορά στην προσέγγιση ε, μικρότερες οικονομίες έναντι μεγαλύτερων μεσαίων οικονομιών. Σε σχέση δηλαδή με το πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και την ερμηνεία του αν θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί ή όχι. Ιδίω ό,τι αφορά καθεστώς πλέον προτιμητέας χώρας, αφρικανικές κτλ. Υπάρχει ένα περιθώριο ερμηνείας και ευελιξίας που θα συνιστούσα να εφαρμόζεται, αλλά θα σταματήσω εδώ, όχι θα σταματήσω εδώ. Όχι, θα σταματήσω και είμαι ελεύθερος στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σούμπερτ, για την παρέμβασή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους μου, βουλευτές οι οποίοι θα ήθελαν το λόγο. Βλέπω ότι πρώτη ή μάλλον ο πρώτος είναι ο κύριος Λίτς. I'm going to speak in German. Γερμανικά θα Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω. Ξεκαθαρίσατε ε, βάσει τα διάφορα υποθέματα τις βασικές προϋποθέσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η φόρος ανάπτυξη και η βιώσιμη. Ε, και ε, εσείς είπατε ίδιος ότι είτε υπάρχουν φόροι στην εξαγωγή είτε όχι, το αν υπάρχουν μάλλον έχει σημασία για την κάθε χώρα. Αλλά το σημαντικότερο είναι η δημιουργία πλούτου, η δημιουργία υπεραξίας και οι θέσει εργασίας, αν υπάρχουν δεν υπάρχουν, για να δημιουργούνται έσοδα. Και επιπλέον προσθέσατε ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα θα πρέπει να έχουμε εκεί όπου υπάρχει υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ξέρετε το μέσο που λέγεται Aid for Trade, δηλαδή αναπτυξιακή συνεργασία ε, ε, έτσι ώστε να προωθείτε το εμπόριο. Για να μπορεί καν να μπαίνει κανείς στο εμπόριο. Και πώς το αξιολογείτε, αν το γνωρίζετε αυτό το μέσο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι σημασία έχει για σας. Και δεύτερον, αυτό τον καιρό συστήνουμε υποεπιτροπή που μόλις αποφασίστηκε για τα έγγραφα του Παναμά, τα περίφημα Panama Papers και τη φοροαποφυγή. Ε, από τη δική σας σκοπιά αυτό σημαίνει τίποτα. Έχετε καμία άποψη, αντίληψη για το θέμα των εγγράφων του ε, Παναμά και τι σημαίνει αυτό για τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη κτλ. Ευχαριστώ. Κύριε ευχαριστώ και εγώ γερμανικά θα μιλήσω. Να βλέπω ότι φοράτε τα ακουστικά σας. Στην εισαγωγή σας είπατε ότι δεν ξέρετε ακόμα τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, γιατί δεν είναι γνωστές αυτές οι καταστάσεις αρκετό καιρό για να μελετηθεί ο αντίκτυπος. Αλλά υπάρχουν κάποιες εθνικές οικονομίες, όπως είναι η Κίνα, γιατί είχατε και ένα παράδειγμα με ορυχία στην Κίνα, έχουν γνωρίσει κάποια ανάπτυξη εδώ και καιρό και η Κίνα είχε πάρα πολύ μεγάλη προστατευτική οικονομία απέναντι στη βιομηχανία της και αναγκάστηκε να τις ανοίξει αφού έγιναν ανταγωνιστικές οικονομίες και οι βιομηχανίες. Και υπάρχουν και άλλες αναδιόμενες εθνικές οικονομίες θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ποιος, προς ποια κατεύθυνση θα εξελιχθεί. Επίσης, το πρώτο που είπατε και συμφωνώ είναι εύκολος τρόπος να αποκομίζει έσοδα το κράτος. Και είναι και ένα επιχείρημα αυτό δικαιολογημένο, γιατί για να στήσουν την οικονομία τους, να τη χτίσουν οι χώρες αυτές χρειάζονται χρήμα. Και αν τους απαγορεύσουμε με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης να το κάνουν, πού θα βρουν λεφτά τότε και από τι θα αντικατασταθεί αυτό. Ε, στην παρουσίασή σας ε, καταλάβαμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις με διαφορετικό αντίκτυπο αναχώρα με το ίδιο μέσο. Τώρα εμεί κάνουμε συμφωνίες εταιρική σχέσης με διάφορες χώρες. Ε, ε, τώρα θα μιλήσουμε για χώρες Ανατολικής Αφρικής, για ΕΠΑ, ε, με το ΣΑΝΤΕΚ, τη Μεσημβρινή Αφρική. Αν κοιτάξω στη ΣΑΝΤΕΚ όμως ε, οι οικονομίες είναι τελείως διαφορετικές των κρατών. Δεν μπορούμε να έχουμε κουστούμι μια συμφωνία προς όλους. Η Νότια Αφρική σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες έχει ισχυρή οικονομία. Τώρα εμείς ερχόμαστε και κάνουμε συμφωνίες με τις χώρες αυτές όπου ξέρω εγώ, απαγορεύονται οι φόροι στην εξαγωγή και χρησιμοποιούμε μία συμφωνία, ένα μέσο για πολλές χώρες που έχουν διαφορετικές πραγματικότητες. Πώς να το ερμηνεύσω αυτό, γιατί το θεωρώ πρόβλημα. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Νόιζερ και μετά στην κυρία. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της μελέτης. Που είναι πολύ περίπλοκη και πολύ θεωρητική βεβαίως. Εγώ θα επιθυμούσα πιο πρακτική ε, παρουσίαση για την Επιτροπή, γιατί εμεί καλούμαστε συγκεκριμένα, όπως είπε και η συνάδελφος Χόιμπουχ, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, που αποφασίζουμε και που συζητάμε να δράσουμε με τρόπο πρακτικό. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να δούμε τι θα κάνουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε αρνητικέ επιπτώσει στι αναπτυσσόμενε χώρε, διότι αυτό που θέλουμε εμεί είναι να υπάρξει θετική ανάπτυξη είπατε ότι σε ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε περισσότερη τεχνική συνεργασία με περισσότερο ανταγωνισμό. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό. Και μετά αναφέρατε το σύστημα hedging, προστασία με τρόπο νομισματικό σχήματα. Μα είναι σε θέση τώρα οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν τέτοια συστήματα στην οικονομία τους. Το τελευταίο δεν μπορώ παρά να το υπογραμμίσω. Χρειάζεται καλύτερη διακυβέρνηση για να βοηθήσουμε κι εμείς να είναι σε θέση η κρατική μηχανή να αναπαράγει το εισόδημα για να μπορούν οι χώρες να αναπτυχθούν μόνες τους και να αναλάβουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας ήδη. Ευχαριστούμε. Κυρία Χάουταλα τώρα, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη μελέτη και την παρουσίαση κύριε Σούμπερτ. Η ερώτησή μου είναι σχεδόν ταυτόσιμη με την ερώτηση του αδελφού Αρνελίτς και αφορά τα μέτρα for Trade. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να εισέλθουν ε, στις αλυσίδες αξίας. Και βλέπω ότι το Διεθνές ε, Κέντρο Εμπορίου σε σχέση με τον ΠΟΕ κάνει πολύ καλή δουλειά. Όπως και ο Σάφος Λίτς, θα ήθελα να ξέρω και εγώ ποια είναι η άποψή σας για τα μέτρα που θεωρείτε ότι θα ήταν ε, θετικά και θα στήριζαν τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο. Αν όχι, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον κάποιο από τους εκπροσώπους επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ζεν Κοβάλ. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και εμείς για τη μελέτη και για την παρουσίαση. Πράγματι το θέμα είναι πολύ πολύπλοκο. Και αν κάποιος διαβάσει τη μελέτη μέχρι τέλους, διαπιστώνει ότι φωτίζει κάποιες πτυχές με ενδιαφέρον τρόπο στο τέλος, υπερβαίνοντας απλουστευτικές συζητήσεις ότι η φόρτη των εξαγωγών είναι καλή ή κακή και σίγουρα θα βοηθά και εμάς να αποφύγουμε, να περιοριστούμε σε μια κοντόθωρη εξέταση του θέματος. Πάντα υπό όρους καλού κακού. Αλλά να δούμε και τι γίνεται μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, στη μελέτη του δόκτωρος Σούμπερτ ε, λέγεται ότι οι περιορισμοί και οι φόροι μακροπρόθεσμα έχουν επιθύμητα αποτελέσματα για τις χώρες που εφαρμόζουν αυτούς τους φόρους, γιατί μπορούν να μειώσουν τα κίνητρα για την προϊόντα να μειώσουν την απασχόληση και να αυξήσουν τις τιμές. Αυτό που ότι λοιπόν πρέπει να πούμε είναι ότι ναι, αυτό είναι ένα ε, εργαλείο πολιτικής και εξορισμού οδηγεί στην ανάπτυξη. Προφανώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, διότι ακριβώς δεν αντιμετωπίζουν απλοϊκά τους φόρους στις εξαγωγές, αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτοί οι φόροι, ότι οι εταίροι μας ήθελαν αυτές τις, ε, αυτούς τους φόρους να τους διατηρήσουν, να μην τους καταργήσουν ούτε να απαγορεύσουν ε, την ισχύ τους, γιατί όχι απλά μόνο να θέλουν να παραμείνουν αυτοί οι φόροι, αλλά παραδείγματο χάρη στην περίπτωση τη Αφρική υπάρχει και τάση να δεσπιστούν και νέοι φόροι, αλλά βέβαια με διαφανή και σαφή κριτήρια που είναι και αντικείμενο διαπραγμάτευση με του εταίρου μα. Αυτή είναι η πολύ σύντομη παρέμβασή μα. Ολοκληρώνω επαναλαμβάνοντα ευχαριστίες μου στον κύριο Σούμπερτ που έχει σε φως σε κάποιες πτυχές και δείχνει και τι προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε στο πλαίσιο των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις, κύριε Σούμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω κάτι πολύ ακαδημαϊκό. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα, αντί να σας απαντήσω απευθείας σε ερωτήσεις σας, που είναι πολύ σημαντικές βέβαια. Και κάτι θέλω να μας πούν. Στη διαδικασία την αναπτυξιακή, στις εμπορικέ σχέσεις, στις σχέσεις γενικά που έχετε με αυτές τις χώρες, τι θέλετε. Θέλετε χώρες αυτές να αναπτυχθούν στο επόμενο επίπεδο, στο επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, αν παράγουν ένα συγκεκριμένο υλικό, το οποίο το εξάγουν και έπειτα το εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν η πρώτη ύλη στο πλαίσιο μιας διαδικασίας και εξειδικευμένα η ευρωπαϊκή βιομηχανία, στον με τις ε, υψηλή τεχνολογία ενέργεια και έχει την, ε, το προβάδισμα. Τι θέλετε, θέλετε πραγματικά μια άλλη χώρα που είναι ένας εμπορικός εταίρος σας να αναπτύξει πολύ, με πολύ φθηνότερο εργατικό δυναμικό την δυνατότητα να φέρει σε πέρα όλη αυτή τη ε, διαδικασία επεξεργασία και να χάσετε εσείς ε, αυτή τη ε, δραστηριότητα και νομίζω είναι ερώτημα θεμητό και πρέπει να τεθεί. Δεν είναι ευχάριστο. Ούτε από ηθικής πλευράς είναι ευτυχές ερώτημα, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί, διότι η επιτυχημένη ανάπτυξη εκεί οδηγεί. Δηλαδή, η βιομηχανία που έχετε εδώ να μετακατασταθεί και να πάει πιο κοντά εκεί που ε, προέρχονται, από εκεί που προέρχονται οι πρώτες ύλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσετε. Τώρα, αν δείτε τη βιομηχανία των μικροτσίπ, ένα κλασικό παράδειγμα, η βιομηχανία μικροτσίπ είχε κέντρο τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη. Και μετά που πήγε, πήγε στην Ασία. Και έπειτα υπήρχε και μεταφορά γνώσης ε, που είχε ως αποτέλεσμα να πάει στην Ασία η όλη αυτή η βιομηχανία, έγινε πιο φθηνό, πιο ε, οικονομικό να κατασκευάζονται τα μικροτσίπ εκεί, άρα έμεναν πίσω είπα, και η Ευρώπη και η Ασία ε, ήταν... Ε, στο, στην πρώτη γραμμή της μεγάλης οικονομικής αυτής ανάπτυξης. Τώρα 20 χρόνια μετά αντιστρέφεται, αναστρέφεται η τάση, επανέρχεται πίσω δηλαδή στη ΣΥΠΑ ή στην Ευρώπη αυτή η τεχνολογία. Αλλά υπάρχουν λόγοι πίσω από αυτό. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίσετε τι θέλετε εσείς πραγματικά και ποιες είναι οι επιπτώσεις ή ποιε θα είναι οι επιπτώσεις της επιτυχίας τουλάχιστον σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και με τομέα. Για το Aid for Trade, φυσικά και το ξέρω, κατά πόσο είναι καλό αυτό είναι, αδιαμφισβήτητα. Όμως, υπάρχουν κάποιοι όροι ε, βαθμοί αιρεσιμότητας. Παραδείγματο χάρη, που αν θα δώσουν περισσότερη ε, βοήθεια σε σχέση με εμπορικέ συμφωνίε, παραδείγματο χάρη. Σε κάποιες περιπτώσεις, δυστυχώ, πραγματικότητα ε, δείχνει ότι άλλο λειτουργεί αλλού. Θα έλθω και στα έγγραφα του Παναμά. Και στα σχετικά που είναι ένα πιο παράξενο θέμα που έχει να κάνει και με τα κρατικά σώδα κτλ. Αναφέρθηκε η Κίνα. Θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα. Φυσικά και θα μπορούσε, γιατί για πολλά θα μπορούσε να είναι παράδειγμα. Για να βάλουμε την Ινδία όμως, και αυτή ως παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για πολύ μεγάλες οικονομίες. Είναι αναπτυσσόμενες, αλλά τεράστιου μεγέθους, ε, έχουν τεράστιους ε, φυσικούς πόρους, είναι πολυπληθέστατες χώρες, Άρα μπορούν να φέρουν και να παράσχουν κεφάλαιο και εργατικό δυναμικό σε πολύ ευρία κλίμακα. Αν οργανωθούν. Και αυτό δεν ισχύει για μικρές αναπτυσσόμενες χώρες ε, γύρω από τον Ισημερινό. Υπάρχουν και άλλοι όροι που επηρεάζουν και άλλες συνθήκες. Υπάρχει το μέγεθος που σίγουρα στην προκειμένη περίπτωση το μέγεθος μετράει σε σχέση με την αποτελεσματικότητα όλων αυτών που συζητάμε. Κίνα όμως ναι πράγματι μπορεί να ε, μας προσφέρει πολλά παραδείγματα και πολλά παραδείγματα μπορεί κανείς να αναφέρει όπως και δεκαετίες θα έλεγα ε, παραδειγμάτων μπορεί να σκεφτεί κανείς. Όμως έχουμε και την Ινδία που δείχνει πως μπορεί κανείς να αναπτυχθεί. Έφτασαν στην οροφή τους και δεν την ξεπέρασαν γιατί δεν άνοιξαν προς τα έξω. Τεχνική συνεργασία που οδηγεί στον ανταγωνισμό. Και τι σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ε, στοιχεία, που, πολλές ενδείξεις και υπάρχουν ε, και προγράμματα από το UNDP, την UNCTAD ε, έχουν χρηματοδοτηθεί, δημιουργηθεί δίκτυα στη διοστεφαντουργία και αλλού, στην ε, Τζαμάικα και σε άλλες χώρες. Με πολύ θετικά αποτελέσματα. και βοηθεί αυτή η τεχνική συνεργασία τις χώρες να βρουν ε, τεχνικούς εταίρους και να εργαστούν ως υπεργολάβοι, για παράδειγμα. Αυτό έγινε με την Ιταλία, στον τομέα των ε, ε, υποδημάτων, της κλωστεφαντουργίας, του δέρματος κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αγορές των futures. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι κάτι μπορεί να κάνει. Τελευταία φορά το τελευταίο ερώτημα μάλλον αφορά τα Panama Papers που μας δείχνουν το κρυφό χρήμα που κυκλοφορεί, τέλος πάντων κρυμμένο στον κόσμο γύρω-γύρω Αν δείτε τα έγγραφα του Παναμά, που από πού εκλάπει αυτό το χρήμα και τα λοιπά. Μεταξύ άλλων και άψεξα, όχι σίγουρα, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Δεν θα είναι χρήματα που κέρδισε κάποιος με τον ιδρώτα του προσώπου του, μπορεί να έχει να κάνει με φόρους στις εξαγωγές ή άλλες ενισχύσεις ή πώληση όπλων, λαθρεμπόριο και πολλά άλλα τέτοια. Αν αρχίσει να σκάβει κανείς, θα ανακαλύψει τεράστια επίπεδα διαφθοράς. Και σίγουρα υπάρχει μεγάλη σχέση με τον αναπτυξιακό κόσμο. Très Ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο μας, κύριο Σούμπερτ, που ήρθε στην σημερινή μας ε, συνεδρίαση για να μας ε, δώσει αυτές τις πληροφορίες. θα σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και του συναδέλφου που παρενέβησαν και εμπλούτησαν ε, αυτή την απογευματινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Προτείνω το επόμενο σημείο 8 τη ημερήσιας διάταξης, εταιρική, συμφωνία εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη τη και τα κράτη και της ε, ΚΑΜΑ και των κρατών ΣΟΕΣ. Όχι, ΣΟΕΣ είναι συμφωνίες α, και συγγνώμη, τα, κράτη της, ε, Ανατολ, της Μεσημβρινής Αφρικής. Πρόκειται για συμφωνία με έξι από τα 15 μέλη της ε, κοινότητας ε, ανάπτυξης της Νότιας Αφρικής, Μποτζουάνα, Λεσότο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη. Αυτή η συμφωνία ε, στηρίζεται στην ανάπτυξη και επιδιώκει το στόχο της ε, οικονομικής ε, περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνυπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή στο Καζάνε της Μπουτσουάνα Και τώρα περιμένουμε, είμαστε μάλλον στη φάση όπου το Συμβούλιο θα πρέπει να έρθει προς το Κοινοβούλιο για να λάβει θέση και γι' αυτό και έχουμε τώρα να ακούσουμε τον εισηγητή μας, Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, είμαστε σήμερα εδώ για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση σε αυτήν ε, την Επιτροπή για το αντικείμενο της γνωμοδότησης για αυτή την ε, συμφωνία εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της και τα κράτη-μέλη της της ΚΑΜΑ, των χωρών δηλαδή της Μεσηβρινής Αφρικής, Βοτζουάνα, Λεσότο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη. Ε, εδώ στις 23 Μαΐου είχαμε ήδη μια πρώτη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Και φυσικά η Επιτροπή Διεθνούς Υπορείου είναι η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, αυτή η συμφωνία υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου, δεν, δεν και λίγες μέρες δηλαδή, αν και οι διαπραγματεύσει ολοκληρώθηκαν πριν από δύο χρόνια σχεδόν, τον Ιούλιο του 2014. Τότε, αυτά τα δύο χρόνια μας φαίνονταν πολύ χρόνος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα είχε ορίσει την 1η Οκτωβρίου ως προθεσμία εντός της οποίας θα έπρεπε να γίνει η κύρωση της συμφωνίας και μάλιστα αυτή η προθεσμία διατηρείται. Διαφορετικά οι χώρες αυτές θα έχαναν τη καθεστώς ε, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω της εφαρμογής των κανόνων του ΠΟΕ. Η συμφωνία αυτή αφορά αποκλειστικά το εμπόριο αγαθών είναι μια, μια ε, αμοιβαία συμφωνία και άρα συμβατή με τους ε, κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορία και χαρακτηρίζεται από την ασύμετρη φύση και τη σταδιακή φύση της. Έρχεται να αντικαταστήσει το καθεστώς πρόσβασης αγοράς για τις χώρες ΑΚΕ που δεν ε, έχουν το καθεστώς των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, δηλαδή το σύστημα των μονομερών προτιμήσεων ώστε αυτά όλα να καταστούν σύμβατα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτό που οφείλει τώρα να κάνει το Κοινοβούλιο σε αυτή τη φάση είναι να λάβει θέση, δηλαδή να εγκρίνει ή όχι αυτή τη συμφωνία. Τη συμφωνία από αυτή που έχει υπογραφεί και που υπογράφηκε μετά από διαπραγματεύσει. Θα πρέπει να τονίσω ότι μέχρι και την περασμένη εβδομάδα στην Αμίμπια, στην Βιντόκα, έγινε συνεδρίαση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, χώρες ΑΚΕ, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, όπου οι αφρικανικές χώρες επανέλαβαν την πολιτική τους βούληση να ολοκληρώσουν αυτή την συμφωνία και να τεθεί σε εφαρμογή αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης κατεπηγόντως. Στο σχέδιο γνωμοδότησης που σας υπέβαλα, υπογράμμισα ότι η συμφωνία αυτή η ασυμμετρική αυτή εταιρική σχέση επιτρέπει στις ε, λόγω αφρικανικές χώρες να προστατέψουν τους ευαίσθητους τομείς ε, παραγωγής τους απέναντι στους ευρωπαίους ανταγωνιστές. Περιλαμβάνει διάφορες ρήτρες ασφαλείας, πέντε τον αριθμό, μέσα στις οποίες ε, η δυνατότητα αυτόματης προστασίας ε, των γεωργικών αγορών ε, και άλλες ρήτες που αφορούν ε, την ασφάλεια προμηθειών σε τρόφιμα. Και επίσης να τονίσω ότι αυτή η συμφωνία επιτρέπει την εξάλληψη της προσφυγής σε επιδοτήσεις στις εξαγωγές για τα αγροτικά προϊόντα που ήταν ένα σημαντικό ζήτημα που αφορούσε τις χώρες της, ε, ε, της ΚΑΜΑ και επίσης περιλαμβάνει κανόνες προέλευσης σχετικά ευέλικτους ε, που σε ειδικέ περιστάσεις μπορεί και μέχρι και να οδηγήσουν στην εφαρμογή φόρων επί των εξαγωγών. Πράγμα που εξάλλου θεωρούμε και σε συζήτηση που κάναμε πρόσφατα εδώ, είπαμε ότι είναι συμβατό τελικά και επιτρέπεται από τις κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Υπάρχει λοιπόν άρθρο σε σχέση με το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη, ρήτρες προστασίας όσον αφορά την εργατική νομοθεσία και την παρεμβαλλοντική νομοθεσία και επίσης ε, προβλέπει διαδικασία διαβούλευσης για τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και ένα κεφάλαιο που αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Ωστόσο θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο πτυχές που είναι πολύ σημαντικές. Καταρχάς πρέπει να εξασφαλίσουμε το αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της διαδικασίας εφαρμογής αυτής της συμφωνίας και αυτή η παρακολούθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εμπλέκει την κοινωνία των πολιτών, αλλά και να κινητοποιεί κατάλληλους πόρους ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα των αφρικανικών χωρών που είναι εταίρημα σε αυτή τη συμφωνία ε, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης ορισμένων, ορισμένου κόστους προσαρμογής που σημαίνει μια τέτοια είδους οικονομική μετάβαση. Ε, Επίσης θα ήθελα να εκφράσω την ε, ε, θλίψη μου, διότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία μια αυτόνομη ρήτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει επανελειμμένως. Ε, αναφορά και αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού και είναι λυπηρό που αυτή η συσχέτιση, η σύνδεση με το καθεστώς πλαίσιο δεν διατηρείται. Θα έπρεπε να διατηρηθεί και πέρα από την ε, ε, χρονολογία ε, εκπνοής της Συμφωνίας του Κοτονού που είναι το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλαμε να μας ενημερώσει για το πότε θα μπορέσει να δημοσιεύσει τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης αντικτύπου της συμφωνίας τούτης. Σε μια πρώτη προκαταρτική μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών ε, λέει πως έχει αυτή η συμφωνία θετικό αντίκτυπο, αλλά περιορισμένο. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε και ένα σχόλιο της Επιτροπής για αυτά τα θέματα. Αλλά το πιο σημαντικό ζήτημα, και με αυτό κλείνω κύριε Πρόεδρε, είναι ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό, σεβαστή προθεσμία για την κύρωση από πλευρά ΑΚΕ. Γιατί εφόσον έχει υπογραφεί στις 10 Ιουνίου, να δούμε ότι οι διαδικασίε κύρωση από πλευρά των κοινοβουλίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή λίγο παραπάνω από τρει μήνε έχουμε στη διάθεσή μα. Είναι λίγο σύντομη αυτή η περίοδο, πολύ σύντομη αυτή η περίοδο. Που παρότι συζητώνται για πολύ χρονικό διάστημα, στα κοινοβούλια τώρα πρέπει να συζητηθεί η συμφωνία και να κυρωθεί. Γι' αυτό και θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να δημιουργήσουν γρήγορα ή να, να λειτουργήσουν μάλλον γρήγορα οι δημοκρατικές διαδικασίες γιατί μας πιέζει ο χρόνος και γι' αυτό και θέλω να επιμείνω σε μια ερώτηση που ήδη έχει διατυπωθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε μήπως αυτή η προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου μπορεί να παραταθεί. Γιατί απαιτεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ένα λογικό χρονικό διάστημα για την κύρωση και εδώ τώρα δεν είναι λογικό αυτό το διάστημα που έχει μείνει. Τώρα, εμείς θα πρέπει ως Επιτροπή Ανάπτυξης να εκφράσουμε τη γνώμη μας και η άποψή μου είναι ότι θα αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να συστήσει στην Ολομέλεια να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Υπογραμμίζοντας αυτές τις πολύ σημαντικές ε, πτυχές, παρακολούθηση, ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης ε, το θέμα των προθεσμιών για την κύρωση της συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ αγαπητέ συνάδελφε. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που το επιθυμούν. Καταρχήν στους σκιώδεις. Πρώτη την κυρία Χόλμποχ. D'accord. Pardon, excusez-moi. Euh, Madame euh, euh, Bouche, je vais passer la parole au collègue euh, Zara Zaradil. Συγγνώμη, κυρία Χολμπούχ, θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ζαχραντήλ. Mm. όχι, όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Θέλω να πω Άνταμ. Mm.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 Μεταρχάς, η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες ε, της ε, κοινότητα, αναπτυξιακής κοινότητας της ε, Νοτιού Αφρικής είναι σημαντικό να μιλήσουμε για αυτή τη συνεργασία, να συστήσουμε θετικά την έγκριση αυτής της συμφωνίας, όχι μόνο προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αλλά και προς το Συμβούλιο ότι δηλαδή θα πρέπει να κυρώσει αυτή τη συμφωνία. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με τους στόχους και την ε, ολοκλήρωση των χωρών αυτών και την ένταξή τους στην παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη πλευρά πρέπει να θυμίσουμε και τα θέματα που σχετίζονται με την βοήθεια της στήριξη που μπορεί και δίνει η πλούσια Ευρώπη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως, να πω επίσης ότι πέρα από αυτές, αυτούς τους ευσεβείς πόθους και τους αξιέπαινους στόχους υπέρ της ανάπτυξης αυτών των χωρών, είμαι πεπισμένος πως η συμφωνία αυτή θα είναι χρήσιμη και για τα δύο μέρη. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Είμαι πεπισμένος ότι στην ε, Ήπειρό μας ε, λίγοι άνθρωποι πιστεύουν ότι, ότι είναι δίκαιο να υπάρχει αυτό, αυτή η διαφορά και αυτή η χάσμα ε, ε, ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, χώρες ε, αλλά και για την ανθρώπινη κατάσταση. Η ανθρώπινη υπόσταση θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να παγκοσμιοποιηθεί το καλό. Σε αυτό χρησιμεύει αυτή η συμφωνία. Επιπλέον να, πω ότι ίσως να έχει κάποια ε, προβλήματα αυτή η συμφωνία, ιδιαίτερα τα, οι προθεσμίες είναι σχετικά μικρές. Και επίση ε, δεν αναφέρονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κοινότητα ανάπτυξης, αναπτυξική κοινότητα της Νότιας Αφρικής δεν έχει να ασχοληθεί μόνο με θέματα ανάπτυξης και εμπορίου, αλλά κυρίως και με θέματα που σχετίζονται με την ε, αξία της ανθρώπινης ζωής, των πολιτικών δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών που θα πρέπει να ανέλθουν στις προδιαγραφές που έχουμε εδώ στην Ευρώπη, στις, ε, στα δικαιώματα που εμείς ε, έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ευρώπη. Γι' αυτό και θα πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγις ώστε η Συμφωνία του Κοτονού να συνεχίσει να υπάρχει σε αυτού του είδους τις συμφωνίες και έτσι ακόμα και μετά την εκπνοή του Κοτονού να συνεχίζεται αυτή η αναπτυξιακή προσπάθεια και να επιστήσω την προσοχή σας κλείνοντας σε ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέρθηκε. Δεν είναι σημαντικό μόνο αυτή η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή. Είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε και την εφαρμογή της, ώστε να δούμε ότι όντως αποφέρει αποτελέσματα. Δεν φτάνει να το υπογράψουμε και μετά το ξεχάσουμε. Θα πρέπει και αυτή η υπογραφή να αποφέρει τους καρπούς που επιθυμούν και οι δύο πλευρές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Ντέβα. Συνάδελφε, παρακαλώ με παρεξηγήσετε, αφού θα πω αυτά που θα πω. Για πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε με τις, τις ε, ε, των διαφόρων ε, συμφωνιών με τις χώρες ε, τις αφρικανικές και έχουμε δώσει πολλή στήριξη και μέσω του EDF. Αλλά κάτι αρχίζει να με ανησυχεί. Χώρες που δεν έχουν πολύ στενές εμπορικές σχέσεις με την Ένωση, όπως οι χώρες του ΑΣΕΑΝ, Καμπότζη και τα λοιπά, έχουν συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μαζί μας. Αλλά αυτές οι χώρες έχουν αναπτυχθεί με ε, αξιοπρόσιτο τρόπο. Και από τη φτώχεια έχουν φτάσει σε χώρες, να είναι χώρες μέσω εισοδήματος και άνω πολύ γρήγορα. Η Κίνα ε, επίσης ε, είναι τώρα η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα χάλιβα στα τελευταία, και αυτό έγινε μέσα στα τελευταία 15-20 χρόνια. Αυτές οι χώρες λοιπόν που δεν, είχαν, δεν βρίσκονταν στις αγκάλες της Ένωσης, ε, που τις κρατούσε δηλαδή έτσι στοργικά, η Ευρώπη έχουν αναπτυχθεί ενώ αντιθέτως αυτές οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση μαζί μας δεν καταφέρνουν να χειραφετηθούν. Η αναπτυξή τους δεν πάει καλά ε, και εμείς εξεκολουθούμε να τους λέμε πώς και τι να κάνουν. Κάτι που τους είπαμε να κάνουμε είναι αυτό το οι, οι, οι συμφωνίες εταιρικής, οικονομικής εταιρικής σχέσης. Μην οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις ε, αλλού. Δηλαδή ελεύθερα συναλλαγές και Τελωνιακή Ένωση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της εκάστοτε ε, εταιρικής σχέσης και κάποιος είπε και μάλιστα ναι και ελεύθερη κυκλοφορία ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Δεν έχουν φτάσει εκεί ακόμα, αλλά μπορεί κιόλα. Το πρόβλημα όμω είναι Οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί αυτών των χωρών έχουν διαμαρτυρηθεί ιδιωτικώ σε μένα ότι όταν του επιβάλλουμε αυτέ τι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών και του λέμε να ανταλλάζουν μεταξύ του ελεύθερα, όπω κάνουμε εμεί με τα δικά μα κάτι μελη τα εισοδήματά του από τους τελωνιακούς δασμούς εξαφανίζονται. Και όταν εξαφανίζονται αυτά τα έσοδα του κράτους, ε, εμφανίζεται μια μεγάλη τρύπα στον προπολογισμό. Ε, εμείς δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε αυτή την τρύπα, ενώ στη θεωρία λέμε μην ανησυχείτε γι' αυτό γιατί η εν οικονομία σας θα αναπτυχθεί. Ξανά μανά λοιπόν μου έχουν ε, επαναλάβει αυτό το πρόβλημα. Πώς θα πληρώσω τους δημόσιους υπαλλήλους εφόσον δεν έχω ε, τελωνιακά εισοδήματα, δασμούς. Δεν ξέρω αν ο κύριος Περέρα μπορεί να είναι σε θέση να μου απαντήσει αυτή την ερώτηση, αν κάποιος από την Κομισιόν έχει την απάντηση σε αυτό μου το ερώτημα. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Χόλμπους. Κυρία Χόλμπους, ευχαριστώ Χόλμπου, για αυτή την τοποθέτηση. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα σημεία κριτικής που ακούσαμε και συμμερίζομαι. Ε, είτε είναι η χρονική στιγμή της υποχρέωσης απελευθέρωσης, ε, τα φορολογικά έσοδα, οι απώλειες αυτών επίσης αναφέρθηκαν, καθώς επίσης και η κοινωνία των πολιτών που έχει συμπεριληφθεί πάρα πολύ λίγο, όπως και τα κοινοβούλια. Ούτε υπάρχει ξεχωριστή ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά λείπουν, τα λέει η γνωμοδότηση και τα επισημαίνει και χαίρομαι πάρα πολύ. Πλην όμω διατηρώ τι επιφυλάξει μου και τι αμφιβολίες μου για τη Συμφωνία Οικονομική Εταιρική σχέση. Πρώτον, ε, η Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αφρική είπε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες ε, υπονομεύουν την περιφερειακή ολοκλήρωση στην Μεσημβρινή Αφρική. Δεν θα πρέπει εμείς αυτό να το επιθυμούμε. Και εδώ και λίγο καιρό γίνονται διαπραγματεύσεις για μια παναφρικανική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών σε όλη την Ήπειρο. Και εκεί πάλι η Οικονομική Επιτροπή για την Αφρική, πάντα των Ηνωμένων Εθνών, συνιστά να ε, ολοκληρωθεί αυτή πριν υπογραφούν οι οι Συμφωνίες Οικονομικής και Εμπορικής σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πριν τεθούν σε ισχύ για να αποφύγουμε τι ανετικές συνέπειε. Και ε, παραμένουν οι αμφιβολίε μου. Νομίζω ότι αυτή η ε, αμοιβαία απελευθέρωση του εμπορίου τόσο νωρίς δεν ξέρω κατά πόσο θα επιφέρει ένα ε, ανθυρό τοπίο στην οικονομία τους. Επαναλαμβάνω, οι χώρες της ε, ε, ΣΑΝΤΕΚ που είναι η κοινότητα ανάπτυξη Νοτιού Αφρικής διαφέρουν οικονομικά. Εκεί κυριαρχεί οικονομικά η Νότια Αφρική σε σχέση με τους γειτονές της και τους επιβάλλεται και φοβάμαι ότι θα έχει αμυντικές συνέπειες ή θα μπορούσαμε να στρέψουμε τη μία χώρα ενάντια στην άλλη αν προχωρήσουμε σε αμοιβαία διάνοιξη των αγορών. Θέλω να θυμίσω εδώ ή να επαναλάβω μια πρόταση που ταιριάζει πάρα πολύ καλά σε σχέση με αυτό που ακούσαμε προηγουμένως για την κατάργηση των φόρων εξαγωγής. Ένα μέλος ΑΚΕ την περασμένη εβδομάδα στη συνεδρίαση είπε το εξής. Χρειάζεται προσοχή εδώ να μην αναπτυσσόμεθα εις το διηνικές και να μην είμαστε για πάντα αναπτυσσόμενες χώρες. Πότε γινόμαστε ανεπτυγμένε, Δηλαδή το θέμα είναι τι θέλουμε πραγματικά, να είμαστε για πάντα αναπτυσσόμενε. εμεί τι θέλουμε, οι χώρε αυτέ να ξεφύγουν από το να είναι εξαγωγή πρώτων υλών και να μπορούν μόνες του να παράγουν ε, προϊόντα μεταποιημένα τα οποία αυτή τη στιγμή εμεί παράγουμε στι χώρε μα Το θέλουμε αυτό και με τις συμφωνίες αυτές οικονομικής εταιρικής σχέσης. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις χώρες αυτές το καθεστώς των προμηθευτών, ορυκτών και πρώτων υλών ή μήπω να μπορούν να τα παράγουν οι ίδιες και τότε η δική μας ανάπτυξη ποια θα είναι. Τότε το κατάλαβα εγώ την περασμένη εβδομάδα, το τάξω όλα αυτά. Και προηγουμένως από τον καθηγητή Σούμπερτ που το έθεσε. Και με αυτές τις συγκεκριμένε συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης δεν έχουμε απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να λάβει τώρα το λόγο η κυρία Σάντρα Γκαλίνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Good afternoon and many thanks for inviting. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συνοδεύομαι κύριε Πρόεδρε και από τον Χαστάλπουλ από τη ΓΑΜΑ έναν συνάδελφο ο οποίος ε, ασχολείται με τις σχετικές συμφωνίες ε, με τη ΣΑΝΤΕΚΑ. Η έκθεση ήταν πολύ ευχάριστο ανάγνωσμα, διότι ε, περιγράψατε με μεγάλη αντικειμενικότητα και ανάλυση την συμφωνία και με τα χαράς διάβασα το έγγραφο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ενδιαφέρον ο διάλογος που έγινε εδώ, γιατί έτσι πήραμε κάπως ε, και μία ιδέα για τις αντιρρήσεις σας, τις ενστάσεις σας. Εγώ θα ήθελα να περάσω στα ερωτήματα και μετά θα κάνω κάποια τελικά ε, σχόλια. Θα απαντήσω μία-μία στις ερωτήσεις, εκτός και αν ξεχάσω καμία που θα μου το θυμίσετε σε ό,τι αφορά την μη εκτελεστική ρήτρα. Εδώ, non-execution ε, clause. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα στη Συμφωνία Κότων. Υπάρχουν όλε οι ρήτρε που μπορείτε να φανταστείτε και κυρώσει που σε άλλε συμφωνίε ε, ελεύθερων συνεργών δεν υπάρχουν. Να έχετε υπόψη λοιπόν ότι σε ε, ΣΟΕΣ έχουμε τηρήσει τα ανώτατα δυνατά πρότυπα. Μίλησαμε για την εκπνοή της Συμφωνίας Κοτονού και εγώ είχα πει ξεκάθαρα ότι οι αρχές ε, που διέπουν τις συμφωνίες αυτές, ακόμη και αν εκπνεύσει η Κοτονού, παραμένουν, άρα οι εταίροι μας έχουν αναγνωρίσει ότι η Ευρώπη πρέπει ε, να ε, παραμείνει και να υποστηρίζει τα ανθρώπινα αυτά δικαιώματα και έχουμε τα συγκεκριμένα μέσα, παρότι μπορεί να εκπνεύσει η Συμφωνία Κοτονού. Ένα άλλο θέμα που ανέκυψε είναι το χρονοδιάγραμμα μικρό, μεγάλο κτλ. Θέλω να διασκεδάσω το φόβο σας για τις χώρες περιοχής. Τρεις χώρες που ε, όχι απλά είναι αποφασμένες, αλλά θέλουν να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατό, έχουν ε, πάει στα κοινοβούλια τους πριν εμείς προχωρήσουμε στην ε, υπογραφή, δηλαδή έλαβε υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, επειδή είχε επιληφθεί ήδη ε, τη συμφωνία, τη εξέταση τη συμφωνία στο Κοινοβούλιο των χωρών αυτών, το λεγόμενο Πρεσεζίν. Και είναι καλό να ε, σας πω ότι τις ε, εξετάσαμε και νομοτεχνικά αυτές τις συμφωνίες η επιλογή των δύο ετών δεν ήταν δική μας επιλογή. Οι εταίροι μας ήθελαν να μελετήσουν το κείμενο από νομικής πλευράς. Και χρειάστηκε χρόνος γι' αυτό, αλλά εγώ προσωπικά είμαι συγκρατημένη αισιόδοξη και ελπίζω να συμφωνήσετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, τα έσοδα από τα εισδασμούς, πολύ καλό το ερώτημα. Πόσο για τους φόρους στις εισαγωγές ούτε 0,6% δεν παίρνουν. 0,59. Ούτε μια ποσοστία μονάδα μείωσης δηλαδή. Βέβαια στην ιστοσελίδα θα αναρτηθεί η μελέτη, το ζήτησε νομίζω ο εισηγητής. Έχουμε ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις μας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα η μελέτη και ακόμη και για τις ε, δημοσιονομικές απώλειες όπως τις ε, ονομάζουμε δεν θα έχουμε πρόβλημα για την περιοχή αυτή. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Κύριος Ντέβα, όχι, όχι, όχι. Αλλά σας χάνω λίγο. Τι είπατε, ένα... Ναι, όμως τα κρατικά έσοδα τι ποσοστό έχουν. Ακόμα μικρότερο είναι η απάντηση. Γιατί μέσα εκεί, αν χάνεις για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση των φόρων από 0,59, καταλαβαίνετε το ποσοστό πόσο είναι. Δεν είναι βέβαια ένα και άκρο προστατευμένο μέσω τη Αφρική αυτό σε σχέση με την Ευρώπη τουλάχιστον. Ίσως είναι η κληρονομιά τη TDCA, αλλά εκεί οι δασμοί δεν είναι ο, φο, τρόπος με τον οποίο κατά ανάγκη ε, χρησιμοποιήθηκε για να προωθηθεί η οικονομία, για να ρυθμίσεις. Δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα εκεί. Είναι όμως μια από τις διατάξεις που έχουμε για όλες τις ε, ΣΟΕΣ και θα επιμείνουμε. Το θέμα είναι εσωτερικό για τη ΣΑΚΟΥ πιο πολύ, γιατί μέρος αυτών των εσόδων αναδιανέμονται μεταξύ των κρατών. Θα πρέπει να αποφασίσουν λοιπόν πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή. Και είναι πολύ λογική και αλληλεγγύη προσέγγιση τους το Λεσότο, για να το πω δηλαδή. Με το όνομά του είναι η χώρα που έχει ένα θέμα, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι και τόσο προβληματικό για την περιοχή εν γέννη. Νομίζω αυτές ήταν οι απαντήσεις που είχα να δώσω. Α, ναι, κοινωνία των πολιτών. Ίσως είναι το πιο σημαντικό. Ετέθη, θα έλεγα, σε σχέση με το γεγονός ότι ίσως να μην έχουμε δομές. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Το άρθρο 4 της συμφωνίας λέει ότι θα έχουμε συμβουλευτικές δομές στο πλαίσιο των συμμετοχικών διαδικασιών των χωρών. Δεν θα επιβάλλουμε ένα μοντέλο, βέβαια. Δεν νομίζω όμως να είναι προβληματικό το θέμα, γιατί έχουμε ασχοληθεί πολύ με το θέμα της παρακολούθησης, του ελέγχου, όχι μόνο για αυτήν τη Συμφωνία Οικονομικής Τερκής, αλλά και για άλλες ο κ. Σάντα νομίζω τα είπε, δεν ε, βάζουμε απλά σταυρού σε τετραγωνίδια, κοιτάμε και την κατάσταση εκ των υστέρων, παρακολουθούμε τα πράγματα για να δούμε αν τα υποσχόμενα ε, με αυτές τις συμφωνίες έχουν εκπληρωθεί και εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά προσιλωμένοι στο στόχο να έχουμε καλή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, της πραγματικής κοινωνίας των πολιτών, δεν κάτι απλό, όπως φαντάζεστε. Και δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, αλλά πραγματικά πρέπει να ζητήσουμε την πραγματική κοινωνία των πολιτών. Πάντως παρακολουθούμε τα πράγματα για να δούμε κατά πόσον ε, οι προσδοκίες που έχουμε για την ανάπτυξη εκπληρώνονται. Αυτές είναι ερωτήσεις μου. Οικονομική υπεροχή ε, και τα λοιπά, Νότιος Αφρική. Οι χώρες αυτές, με βάση τις προσφορές, έλαβαν κάποιες αποφάσεις και στο πλαίσιο μιας ε, επίπονης ε, μακράς διαδικασίας. Και έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία είναι για αυτές σημαντικά κατάντη θα έλεγα. Δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με προσθέμενη αξία, τα προστατεύουν, τα θωρακίζουν και πολύ σωστά κάνουν και καλά κάνουν. Γιατί θέλουμε να σπάσουμε τον κύκλο των πρωτολών και θέλουμε οι χώρες ε, να έχουν περισσότερη προστέμενη αξία στις εξαγωγές τους. Ε, συμφωνείτε μαζί μου, αυτή είναι και μια περιφερειακή τους, αν θέλετε, φιλοδοξία, γιατί πράγματι εν μέρη κυριαρχεί η Νότια Αφρική σε αυτή την περιοχή, αλλά είναι και η ατμομηχανή, ε, ο μοχλός. Κάτι που είχαμε ακούσει από πολλούς υπουργού όταν δεν παραδευόμασταν τη συμφωνία, έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει το που γίνεται η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, αλλά και να συμμετέχουμε στην παραγωγή. Ε, μία αλυσίδα παραγωγή αξίας στην περιοχή. Άρα αυτό που είναι σημαντικό για τι χώρε στη συμφωνία αυτή είναι οι κανόνες προέλευση. Λίγο πολύ ότι ισχύει και για την άλλη συμφωνία που θα συζητήσετε στη συνέχεια. Οι κανόνες προέλευση που θα επιτρέπουν τη σώρευση και όχι μόνο σώρευση με τις χώρες της περιοχή, αλλά και με άλλους δικαιούχους ε, ΣΟΕΣ. Πολύ καινοτόμο αυτό και με τις άλλες ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών γενικευμένων προτιμήσεων. Είναι κάτι νεοτεριστικό για να βγούμε από αυτόν τον κύκλο των πρώτων λόγων κτλ. Είχαμε ένα Ιντερλούδιο μουσικό. Ναι, ωραίο ήταν. Διασκέδασα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι είμαι και πολύ ευγνώμων προς τον εισηγητή που είπε ότι θα δώσει σύμφωνη γνώμη, διότι πράγματι πολύ χρόνος και πολύ νερό έχει πέσει στο μήλο. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε εδώ και την Νότια Αφρική. Θέλουμε πραγματικά να έρθει σε, να υπάρξει ένα αίσιο πέρας σε όλη αυτή την ιστορία, ένα happy end. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μα, όλου του συναντέλφου ε, για την υποστήριξή του για αυτή τη συμφωνία. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να προσθέσει κάτι ο συνάδελφο για την υποστήριξη. Νομίζω όμω ότι σημειώνουμε ότι χρειάζεται να υπάρξει υποστήριξη και μάλιστα κατάλληλη υποστήριξη για όχι μόνο για αυτή την ΣΟΕΣ αλλά και για όλε τι σχετικέ συμφωνίε. Um, um, Όπω ξέρετε, έχουμε σχέδιο να συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας στην Αφρική. 70 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην Αφρική προβλέπονται με τον ιδιωτικό τομέα. Με μόχλευση 4,8 δις θα γίνουν 60. Ε, αυτά τα λεφτά πού θα πάνε αν ε, ε, προχωράμε μόνο σε εξόριξη ε, ορυκτών και πρώτων υλών για να τα στείλουμε στην Ευρώπη, όπως έχουμε κάνει τα τελευταία 150 χρόνια και προς τη θέμενη αξία και ο πλούτος παράγεται εδώ στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στη Βρετανία, τότε ό,τι επενδύσεις και να κάνεις σε εταιρική σχέση, σε ΣΔΙΤ, με το δημόσιο τομέα δεν θα πιάνουν τόπο. Τι θα γίνει, όλες τα τρόφιμα τα φρέσκα λαχανικά, τα, ε, το κρέας, όλα αυτά τα εξάγουμε προς εκεί. Ε, και, εξάγουν εκείνοι ε, πρώτες ύλες και τρόφιμα ε, χωρίς να τα επεξεργάζονται και να τα μεταποιούν. Δηλαδή, τι θα, θα πάνε σε κονσερβοποιίες, θα πάνε σε εργοστάσια, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, αυτό ρωτάω και θα ε, παραχθεί πλούτος για την Αφρική η οικονομία με επενδύσεις εκεί. Γιατί εμείς πάμε εκεί και τους λέμε δύο επενδύσεις και τους παίρνουμε τις πρώτες σύλλες. Πώς το βλέπετε αυτό. Hemstout από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ προφανώς ακόμα δεν έχουμε τις λεπτομέρειες της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής βέβαια στην ανακοίνωση αυτή. Ε, βεβαίως τα χρήματα ε, θα στραφούν στον ιδιωτικό τομέα σε ε, αυτές τις δραστηριότητε στις οποίες υπενήσεστε, αλλά τα χρήματα αυτά δεν είναι μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, είναι για υποδομές ε, και ένα χαρμάνι ολόκληρο. Είναι συνολικό πακέτο, αλλά θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να δούμε τη συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει δεσμευθεί να έρθει μέσα σε ένα τρίμηνο. Η φιλοσοφία είναι ακριβώς αυτό να κινητοποιηθεί στην Ευρώπη ο ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να συμμετέχει σύμφωνα με την ε, ατζέντα της Αντισαπέμπα για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Όχι μόνο για το ιδιωτικό αλλά και ΕΣΔΙΤ και για ε, δημόσιες επενδύσεις κανονικές κρατικές. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την πρόταση. Ναι, επειδή είμαστε πολύ κοντά ε, ε, στη φάση προκήρυξης και τις χώρες έχουμε αρχίσει να συζητούμε τις στρατηγικές ε, ΣΟΕΣ εφαρμογή. Η Μποτσουάν, ας πούμε, έχει τεράστιο δυναμικό στον αγροδιατροφικό τομέα. Θα πρέπει να δούμε τα θέματα του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων που καμιά φορά αγγίζουν στις υποδομές. Ξέρετε ότι εκεί έχουν βουβάλια έχουν σε μια άγρια κατάσταση να βόσκουν σε τεράστιες εκτάσεις. Δηλαδή οι χώρες αυτές δεν εξαγούν μόνο ε, μεταλλεύματα, εμπορεύματα ή ακόμα και ξέρω εγώ κονσέρβες. Δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Ας πούμε, εκεί έχουν ζαχαροκάλαμο, μπορούν να έχουν κονσερβοποιίες και να παράγουν κονσέρβες φρούτων, ε, αντί να εξάγουν τα φρούτα και να τα συσκευάζουμε στην Ευρώπη. Δεν θέλουν τη βοήθεια για τη βοήθεια, ελεημοσύνη. Θέλουν ένα συγκεκριμένο είδος παραγωγής. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβράβευση και ανταμοιβή. Έγινε ε, αναφορά σε τι ε, ανάπτυξη θέλουμε, ποιες ήταν οι φιλοδοξίες της Ασίας και πώς υλοποιούνται ή τα οράματα της Αφρικής και πώς όλα αυτά τα χρόνια έχουν εξατμιστεί, εξανεμιστεί ή ε, καταστραφεί. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και υποδείγματος. Όπως έλεγε ο Πεσπασιανός, Πεκούνιανο Νόλετ, εάν θέλουν να έρθουν οι Κινέζες, επενδύσουν στην Αφρική, χωράνε όλοι. Η Ήπειρος αυτή έχει πολύ λίγες υποδομές σε σχέση με τις ανάγκες είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Καλώ να ορίσουν και καλώς να ορίσει ο ευρωπαϊκός δημόσιος τομέας, ε, συγγνώμη, Αυτά είναι τα πλέον εκτίματα που μπορεί κανεί να έχει στι χώρες αυτές. Δεν είναι μόνο η γενεοδορία ε, του εργατικού δυναμικού, αλλά έχουν και πολύ καλές προτεσίλε που μπορούν να επεξεργαστούν εκεί. Αν ενδιαφέρεστε μπορούμε να σας δώσουμε και λεπτομέρειες και να το συζητήσουμε λεπτομέρως, αλλά ήδη συζητούμε στρατηγικέ εφαρμογής από χώρα σε χώρα, αναχώρα δηλαδή. Ευχαριστώ. Euh, Θα δώσω το λόγο στο συντάκτη ομοδότηση για να κλείσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και για τα σχόλια και για τις ε, προτάσεις όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις της. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κοινοβούλιο μας να δούμε ε, την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πόσο δεσμευμένη είναι ε, στον έλεγχο αυτής της διαδικασίας, έτσι, τον ουσιαστικό και βεβαίως πώς θέλουν να βοηθήσουν τις οικονομίες αυτών των χωρών υπέρ της ανάπτυξης. Και βέβαια μας ενδιαφέρει και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρθηκαν. Um, us... Διότι αυτό είναι ακόμα ε, μεγαλύτερη ε, σιγουριά για μας και άνεση ότι ε, δεν θα λήξει η συμφωνία κοτονού χωρίς να αντικατασταθεί από κάτι άλλο και να υπάρχει νομικό κενό. Ε, μας καθισχάζει αυτό δηλαδή. Ε, να απαντήσω σε κάποια θέματα. Κάποιος συνάδελφος αναφέρθηκε σε αυτά. Δεν θα έλεγα ότι χώρες αυτές που δεν έχουν εμπορική σχέση με την Ευρώπη τα πάνε καλά, ενώ οι υπόλοιπες τις έχουμε καταστρέψει και επικρατεί μεγάλη φτώχεια και δυστυχία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού με το γεγονό αυτό. Η Κίνα, για παράδειγμα, που ακούσαμε προηγουμένως για την ανάπτυξή της, ε, και μπήκε και πιο γρήγορα στον ΠΟΕ και εντάχθηκε στην παγκόσμια οικονομία εκείνα καλύτερα. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι αυτές οι ΣΟΕΣ συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης δεν είναι και η σούπερ επιλογή. Μια συμφωνία είναι. Οι συμφωνίες πάντα είναι επιλογές. Αλλά εδώ ε, εντασσόμεθα και υπακούμε στους κανόνες του ΠΟΕ. Και αν υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς ε, χωρών ε, και και ιδιαίτερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες να προχωρούν σε αυτές τις συμφωνίες, ε, το ξέρουν ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους κανόνες του ΠΟΕ ε, αν δεν υπάρξουν αυτές οι συμφωνίες. Οι παλιοί κανόνες δεν μπορούν να ισχύσουν γιατί δεν έχουν το καθεστώς πια ορισμένες των λιγότερων επιτυγμένων χωρών. Επίσης, η επιλογή που έχουμε εδώ να κάνουμε δεν είναι ακριβώς ε, μεταξύ προστατευτισμού και απελευθέρωση ελευθέρω εμπορίου, γιατί είναι ασύμμετρη η φύση των οικονομιών και των συμφωνιών. Και αυτό δείχνει ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται για απελευθέρωση. Αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε εάν η μεταβατική περίοδος είναι επαρκής ε, λόγω της κατάστασης της κάθε χώρα, μα γι' αυτό χρειάζεται ο έλεγχος και γι' αυτό μπήκαν και οι ασφαλιστικές δικλίδες. Με έναν τρόπο νομίζω ικανοποιητικό. Αυτά. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να κάνω τελικό σχόλιο λέγοντας ότι κατανοώ το επιχείρημα που λέγει ότι χρειάστηκε πολύ χρόνος για να μελετηθούν τα νομικά ζητήματα και αυτά. Εντάξει, ωραία. Τώρα βρισκόμαστε όμως σε μια νέα φάση της διαδικασίας που δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με τις κυβερνήσεις αλλά με τα κοινοβούλια. Δηλαδή καλούνται να κυρώσουν τις συμφωνίες αυτές τα κοινοβούλια. Και αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατική διαδικασία και στις χώρες της Αφρικής, καλό θα ήταν να είμαστε λιγότερο αυστηροί ως προς το χρονοδιάγραμμα, γιατί πρέπει να κυρωθούν αυτά από τα κοινοβούλια τους. Και αυτό θα σήμαινε και ε, ανοιχτή δημοκρατική συζήτηση τώρα ε, στις ε, χώρες αυτές, στα κοινοβούλια τους δηλαδή. Γενικώ ε, φρονώ ότι είναι θετικές αυτές οι συμφωνίες για όλα τα ενεχόμενα μέρη και σας συνιστώ την έγκρισή τους. Κλείνω λέγοντας κάτι στα πορτογαλικά και πάλι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι Ήθελα να κλείσω στα πορτογαλικά για να πω ότι με μεγάλη χαρά βλέπω ότι οι ανεπτυγμένες χώρες προχωρούν και στις χώρες αυτές συμμετέχουν χώρες που μιλούν πορτογαλικά, η Μοζαμβίκη και η Αγκόλα, ελπίζω στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 22 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Και θυμίζω ότι μόνο οι τροπολογίες που ζητούν απόρριψη της σύστασης ε, του εισηγητή είναι παραδεκτές. Η Επιτροπή μας θα ψηφίσει ε, στις 12 Ιουλίου το θέμα αυτό. Βεβαίως, αν στο μεταξύ έχουμε λάβει την επίσημη επιστολή του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και περνούμε στο σημείο 9. Ε, συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών ε, εταίρων της κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής, ΚΑΑ, αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών της Αφετέρου. Ανταλλαγή απόψεων για ίδια συμφωνία που χρειάζεται έγκριση του Κοινοβουλίου και αφορά πλέον τις χώρες κοινότητας Ανατολικής Αφρικής. Πέντε χώρες, Μπουρούντι, Κένια, Ρουάντα, Τανζανία και Ουγγάντα. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν ε, την αναπτυξιακή συνεργασία και το εμπόριο των αγαθών. Ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2014 συντάξει νομοδότησή μας προ ε, προς την Επιτροπή ΙΝΤΑ. Είναι ο συνάδελφος Κριστιαν Πρέντα, στον οποίο διαμέσω λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε μια πληροφορία, ένα νέο που κυκλοφόρησε σήμερα. Το Συμβούλιο σήμερα το πρωί ενέκρινε την υπογραφή της προσωρινής αφαρμογής της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με την κοινότητα των χωρών Ανατολικής Αφρικής. Είχαν ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014 οι διαπραγματεύσεις η συμφωνία είχε μονογραφηθεί δύο μέρες αργότερα Οκτώβριο στις Βρυξέλλες μετά από 12 χρόνια διαπραγματεύσεων. Δεν ήταν και, και λίγα. Σήμερα, επομένως, ολοκληρώνεται μία μακρά πολύπλοκη διαδικασία. Και βέβαια, αυτό που τώρα απομένει να γίνει είναι υπογραφή ε, να δούμε πότε θα οριστεί η ημερομηνία. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έγκριση, ε, σύμφωνη γνώμη, έχει ξεκινήσει το Κοινοβούλιο και όπω είπατε, ανέλαβα τη σύνταξη τη γνωμοδότηση εκ μέρου τη Επιτροπή μα απέναντι στην Επιτροπή τα που είναι καθήλυνα αρμόδια. Εν συνεχεία, το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, Τέσσερις χώρες αφορά αυτή η συμφωνία, Μπουρούντι, Ρουάντα, Τανζανία, Ουγγάντα, δεν και τόσο προχωρημένες και μία έχει μέσο χαμηλό εισόδημα, Κένια. Για τις τέσσερις λιγότερο προχωρημένες, προηγμένες χώρες πρέπει να πούμε ότι ήδη είναι δικαιούχες του καθεστώς ε, όλα εκτός από όπλα, πρόσβαση δηλαδή στις ευρωπαϊκές αγορές ε, με απαλλαγή από ποσοστώσεις ε, και φόρους. Από την άλλη πλευρά η Κένια αυτή τη στιγμή καλύπτεται και μέχρι την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος από τον κανονισμό πρόσβασης στις αγορές και μετά την ημερομηνία αυτή, δηλαδή μετά από 1η Οκτωβρίου 2016 η Κένια θα μπει στο καθεστώς το λιγότερο ευνοημένο των ε, γενικευμένων προτιμήσεων. Με αυτή τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, οι πέντε χώρες της κοινότητας ε, των χώρων Ανατολικής Αφρικής θα έχουν πλέον ένα ενιαίο, μειόμορφο καθεστώς ε, σχέσεων, εμπορικών σχέσεων με την Ευρώπη. Να πω μια λέξη για την κοινότητα κρατών Ανατολικής Αφρικής. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο παράδειγμα ε, που αφορά την Αφρικανική Ήπειρο. Γιατί δεν μιλάμε για μια ενισχυμένη περιφερειακή και οικονομική ολοκλήρωση, θα έλεγα εγώ τελωνιακή ένωση, η οποία είναι επιχειρησιακή από το 2005, αλλά εφαρμόζεται στην πράξη από το 2010 και μετά ακολούθησε η κοινή αγορά το 2010 και η νομισματική ένωση όπως ε, προβλέπεται από το πρωτόκολλο που υπεγράφει το 2013. Έχουμε λοιπόν οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά έχουμε και τη φιλοδοξία δημιουργίας μιας πολιτικής ένωση, Ομοσπονδία Ανατολικής Αφρικής. Το 2013 προβλεπόταν ημερομηνία ε, ολοκλήρωση ε, των εργασιών. Δεν τηρήθηκε η ημερομηνία αυτή για τη δημιουργία μια πολιτική Ένωση, αλλά έχει υπάρξει σε ό,τι αφορά, Πώ να το πω, ε, τα θεμέλια για μια ενδεχόμενη ομοσπονδία. Ο δυναμισμός της κοινότητας των χωρών Ανατολικής Αφρικής έχει εμφανίσει και προσπάθειες προς την υλοποίηση του πλέον φιλόδοξου εμπορικού σχεδίου στην Αφρικανική Ήπειρο. Μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μια τριμερή ζώνη των αλλαγών συγκεκριμένα. Πρέπει να σα πω επίση ότι και το Νότιο Σουδάν έχει προσχωρήσει στην κοινότητα χωρών Ανατολική Αφρική από τη 15η Απριλίου. Και η Σομαλία έχει ζητήσει επίσης να προσχωρήσει. Το δικό μας κοινοβούλιο ήδη και επανειλημμένω έχει πει ότι οι ΣΟΕ, Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, πρέπει να διέπονται από τις ανάγκες των χωρών εταίρων. Και οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει να ευνοούν την ανάπτυξη, την οικονομική διαφοροποίηση, την περιφερειακή ολοκλήρωση, αλλά να συμβάλλουν και στην εκρίζωση της φτώχειας αφετέρου. Και αυτή είναι η στόχη μας, αυτές είναι οι φιλοδοξίες μας που έχουν επαναλάβει πιστάκης. Βέβαια, επειδή πρόκειται για ε, φιλοδοξίες και πολύ φιλόδοξους στόχους. Έχει ξεκινήσει ε, συζήτηση, κρίζωση φτώχειας, περιφερειακή ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι φιλοδοξίες σημαντικές. Έγινε λοιπόν η συζήτηση, θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση με βέβαιος. Περιμένουμε να έχουμε και σήμερα μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Ωστόσο, πιστεύω και θέλω να το αναφέρω, ότι πρέπει τις συμφωνίες οικονομικές εταιρικής σχέσης ναι με να τις κρίνουμε με γνώμονα αυτά τα κριτήρια, αλλά είναι αναγκαίο ταυτόχρονα να αναλύουμε την κάθε συμφωνία με βάση τα δικά της ε, υπέρ και κατά με νυφάλιο τρόπο ή δυνατόν, χωρίς ε, ιδεασμούς. Και καλό θα ήταν να αποφύγουμε να εμπλακούμε σε συζητήσεις που δεν θα οδηγήσουν πουθενά τελικά. Δηλαδή σχέση μεταξύ απελευθέρωσης συναλλαγών και ανάπτυξης. Υπάρχει μεγάλος πειρασμό, ε, η συζήτηση να στραφεί σε αυτά τα μονοπάτια και όχι να κρίνουμε την κάθε συμφωνία με βάση την αξία της. Τα πλονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Να αναφερθώ σε κάποιε λεπτομέρειε, Βέβαια, επειδή μιλάμε ε, για ανταλλαγή απόψεων, χωρίς νομοδότηση, πριν δηλαδή διανεμηθεί κάποιο έγγραφο, δεν το έχουμε ακόμη αποφασίσει. Το σκεφτόμαστε ακόμα. Να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες, κάποια ε, έτσι, προεξέχοντα σημεία να τονίσω. Πρώτον, η συμφωνία αυτή αφορά μόνο προϊόντα. Άρα δεν περιλαμβάνονται οι επενδύσεις ούτε οι υπηρεσίες. Μόνο τα προϊόντα Επίσης, η συμφωνία βασίζεται σε ένα καθεστώς ασύμετρης πρόσβασης. Τι θα πει αυτό η Ένωση, ανοίγει 100% τις αγορές της, όμως οι χώρες της ΚΑ το κάνουν μόνο με ορίζοντα το 2033, δηλαδή σε 17 χρόνια από τώρα. 82,6% σε ό,τι αφορά την αξία των συναλλαγών μεταξύ δύο, των δύο μπλοκ. Οι αγορές τώρα, ε, επειδή ανήκουν οι χώρες στην κοινότητα των χώρων της Ανατολικής Αφρικής, ήδη έχουν ανοίξει επίπεδο 65% και 17,4% των πιο ευαίσθητων προϊόντων αποκλείονται, εξαιρούνται της απελευθέρωση αυτής. Κυρίως γεωργικά προϊόντα, είναι αλκοόλ και άλλα αλκοολούχα ποτά, χημικά προϊόντα, πλαστικό, χαρτί, υφάσματα είδη ένδυσης, υπόδησης, ε, κεραμικά, γυαλικά, οχήματα κτλ. Δεν είναι και λίγα. Η μακρά μεταβατική περίοδος, η το μη επαρκές άγνωσης αγοράς, οι ρήτρες διασφάλισης ε, για τις ε, νεοφυείς ε, βιομηχανίες ε, και τα σχετικά με την επιστηστική ασφάλεια είναι θετικές πτυχές. Από την άλλη πλευρά υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν νέοι προσωρινοί φόροι στις εξαγωγές. Αυτό νομίζω ότι ε, συνιστούν μια ευελιξία και αφήνει και κάποια πολιτικά περιθώρια λιγμών για τους εταίρους. Έχουμε και τις διατάξεις για τους κανόνες προέλευσης που έχουν βελτιωθεί και βελτιώνουν, διευκολύνουν μάλλον τις εξαγωγές και προωθούν την περιφερειακή ολοκλήρωση. 73 σελίδες ε, περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, 21 σελίδες από αυτές αφορούν ε, τα κεφάλαια για την οικονομική συνεργασία και τη συνεργασία για την ανάπτυξη. Αυτό είναι το ε, πολύ βασικό κομμάτι της συμφωνίας. Δεν κρίνεται βέβαια από το μέγεθος μόνο το επιχείρημα, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν, μάλλον όλα θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή, τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας. Και έρχομαι σε αυτό αμέσω. Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από τους οικονομικούς πόρους. Πρέπει να διαπιστώσουμε πάντως ότι υπάρχει πραγματική βούληση να ληφθεί υπόψη ο άξονας ανάπτυξη και να α, ληφθούν υπόψη προκλήσεις που συνεπάγεται για τους εταίρους ε, η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Δεν υπάρχει όμως αναφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Γίνεται απλά μια παραπομπή συμφωνία του Κοτονού. Και αυτό είναι πιο προβληματικό γιατί υπάρχει και η λεγόμενη ραντεβού κλώζ. Δηλαδή θα υπάρξουν ε, συνομιλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και σχετικά και συμφωνία όταν ε, έχουν πέρασει πέντε χρόνια από την εφαρμογή, ε, την έναρξη ισχύω τη συμφωνία. Η βιώσιμη ανάπτυξη, η ρητό, είναι μία από τι παραμέτρου που θα πρέπει να παρακολουθείτε από την Επιτροπή Ανώτατων Αξιωματούχων που θα εποπτεύει την εφαρμογή τη Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση. Αντίθετα με αυτό που ζητούσε το Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει ρήτρα ανθρώπινων δικαιωμάτων και σχετικό αποπτικό μηχανισμό. Ναι, μην υπάρχει ρητή μνήμα στην πρόθεση τη χρηστή διακυβέρνηση. Αυτή είναι η διατύπωση, είναι πιο ευρεία και πιο ασαφή κατ' εμέ, θα πρόσθετα. Επίση, και αυτό θετικό, υπάρχει έμεση αναφορά στο κεκτημένο του Κοτονού ω βάση συμφωνία συμφωνίας, άρθρο 4. Και μιλάμε και για τη ρήτρα Πασαρέλα, άρθρο 136. Τα, μέτρα, τα συμβαλόμενα μέρη μπορούν να πάρουν τα απαιτούμενα με τα δυνάμει των συμφώνων Κοτονού. Βέβαια, γίνεται το ζήτημα μεταξύ του τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία και τη σχέση με τη συμφωνία και τη μετά κοτονού εποχή. Ελπίζουμε να διατηρηθεί η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ενισχυθεί κιόλα στο μέλλον. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα είναι σε ποιο βαθμό ο γενικό μηχανισμό ρύθμισης των διαφορών που προβλέπεται στις ΟΕΣ θα δώσει δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να την εφαρμόσει και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως εδώ θα μπορούσε να μας διαφωτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, δύο σημεία. Πολύ σημαντικά. Το πρώτο, χρηματοδότηση και το δεύτερο, δομές για την υλοποίηση την παραγωγή τη υλοποίηση. Ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, υπάρχει δέσμευση τη Ένωση να εξασφαλίσει κάποιους ε, πόρους ε, με βάση προβλέψεις, αλλά δεν προβλέπονται πρόσθετα κονδύλια. Δηλαδή, υπάρχει ιδέα της προβλεψιμότητας, αλλά όχι πρόσθετα κονδύλια. Τώρα, έχουμε ένα εγγραφό το, της ε, ΚΑ που ορίζει προτεραιότητες και προσδιορίζει τι συγκεκριμένε ανάγκε των χωρών. Αυτά στο πλαίσιο τη εφαρμογή συμφωνία. Θα ήθελα να μα πει η Κομισιόν τώρα ποια είναι τα διαθέσιμα ποσά. Κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν προβλέπεται σε αυτή τη Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση. Αντίθετα με ό,τι ζήτησε το Κοινοβούλιο. Όμω υπάρχει μια κοινή γνωμοδοτική επιτροπή ώστε η κοινότητα των πολιτών να συμμετέχει μαζί με άλλα συμβαλόμενα μέρη και να εξασφαλίζεται έτσι η διάθεση επαρκών πόρων για την κοινότητα των πολιτών. Ένα κατακλείδη, που είναι και προσωρινή η κατακλείδα, γιατί αφού είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και δεν έχουμε και έγγραφο, σίγουρα θα συζητήσουμε εκ νέου το θέμα. Επομένως, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η Συμφωνία Οικονομικής Σχέσης είναι η αρχή και μόνο και η εφαρμογή τη θα επιτρέψει να δούμε κατά πόσον συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη των χωρών ΚΑ και στις ευρύ, μεταρρυθμίσεις ευρεία Ε, είναι αναγκαίο να έχουμε προβλέψει και τους κατάλληλους μηχανισμούς για την εφαρμογή της συμφωνίας. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι δεν πρέπει ε, να παραβλέψουμε τη σημασία που έχει αυτή η συμφωνία ως καταλήτη για εξελίξη στην περιοχή και πρέπει να την προωθήσουμε. Αυτά είναι η δική μου εισαγωγή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Ξεκινάμε με τον κύριο Νόιζερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ τον Κρίστιαν Πρέντα που μας παρουσίασε λεπτομέρως και εξαντλητικός ε, το τι περιλαμβάνουν οι ε, συμφωνίες αυτές με την κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής. Εδώ τώρα έχουμε μια ιδιάζουσα κατάσταση. Έχουμε ολοκληρωμένη τελωνιακή ένωση και νομισματική ένωση ε, στον τομέα αυτό, στη γεωγραφική αυτή περιφέρεια της Αφρικής και το Μπουρούντι, Ρουάντα, Τανζανία, Κένια και Ουγγάντα είναι όλο και περισσότερο ε, ενιαίες στην ανάπτυξή τους στην περιοχή. Και καλά έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντέδρασε στο κοινό τους έτοιμα μείωση των δασμών και το δέχτηκε. Και μέχρι το 2033 θα πρέπει να έχουν ανοίξει αγορές τους κατά το 80% αλλά παραμένει ασύμετρη η συμφωνία αυτή. Λοιπόν, καλά κάναμε και έχουμε και 25 χρόνια στη διάθεσή μας να προετοιμαστούμε. Οι μέχρι τώρα συμφωνίες ήταν ήδη πολύ ανοιχτές και μάλιστα αυτό αφορούσε το ποσοστό του 65%. Δηλαδή ήταν ήδη ανοιχτή η ανάπτυξη. Έχουμε εμείς το εξή σημείο κριτικής τώρα. Όπως είπε και ο Κριστιαν Πρέντα προηγουμένως, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται υπόψη, ούτε τα ε, ε, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν αναφέρονται στις ΣΟΕΣ. Ξέρω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια έμεση μόνο αναφορά στο Κοτονού, αυτή που συμπεριλαμβάνεται, στη Συμφωνία Κοτονού δηλαδή, και μια δήλωση προθέσεων. Πέρα λοιπόν από τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα ότι καταρχήν θέλουμε δεσμευτικές ρήτρες και προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά, τίθεται και ένα θέμα νομικό. Τι θα γίνει μετά την εκπνοή της Συμφωνίας Κοτονού. Συγκεκριμένα, τι θα συμβεί. Γι' αυτό θα μας ενδιαφέρε επιπλέον αυτό να κατοχυρώνεται στη Συμφωνία και ε, θα το προτιμούσαμε. Επίσης, για μας είναι πολύ σημαντικό η εφαρμογή των ΣΟΕΣ να παρακολουθείτε πολύ στενά για να προβλέψουμε και να διορθώσουμε νωρίς ε, στρεβλώσεις και προβλήματα για τις πέντε αυτές χώρες. Κάτι που είναι θετικό είναι ε, ότι προβλέπεται ένα συμβουλευτικό όργανο το οποίο θα συσταθεί, ε, μια συμβουλευτική επιτροπή, Consultative ε, Committee λέγεται αυτό, ε, και να συμμετέχει πολύ καλά η κοινωνία των πολιτών και να παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή και της παρακολούθησης και της εφαρμογής. Λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης στο Μπουρούντι θα πρέπει να προσέξουμε να μην αναβαθμιστεί το καθεστώς μέσω των ΣΟΕΣ αυτών. Ε, βρισκόμαστε σε διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον Μπουρούντι Οπότε στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ε, μας διέπει μια συγκρατημένη έτσι, στάση. Αυτά. Σας είπα, ο Κριστιαν Πρέδα ήταν εξαντλητικός. Θα κάνουμε τις προτάσεις μας και εμείς. Ευχαριστώ πολύ για τη γνωμοδότηση αυτή. Mm, ε, και ε, θα παρακολουθούμε αυτό το θέμα και ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε και από κάποιο διαφορετικό πρίσμα σε σχέση με τις υπόλοιπε ώρες. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ο κύριος Ντέβα. Σας ευχαριστώ. Όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θέλω να ευχαριστήσω τον Κρίστιαν για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Έχω ένα πρόβλημα. <laughs> Για όλη αυτή την υπόθεση. Ξέρουμε ότι η Αφρική μαστίζεται από τη διαφθορά, ολόκληρη η Αφρική. Ξέρουμε ότι γύρω στα ένα τρισεκατομμύριο χρήματα βγαίνουν στα μαύρα από την Αφρική το χρόνο και φτάνουν στις τραπεζές μας και τις ελβετικές τράπεζες. Τι κάνουμε τώρα εμείς, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς τι κάνουμε για τη διαφθορά. Και τι κάνουμε για να εμποδίσουμε να φτάσουν αυτά τα χρήματα που βγαίνουν παράνομα από την, από την Αφρικανική Ήπειρο και πώς ελέγχουμε αυτή τη ροή χρημάτων. Ο συνάδελφος Περέρα έλεγε πριν ότι τα κοινοβούλια αυτών των χωρών θα πρέπει να έχουν το χρόνο να εξετάσουν αυτές τις συμφωνίες ώστε τα οι βουλευτές να μπορούν να εγκρίνουν αυτά τα θέματα. Μα τα κοινοβούλια αυτών των χωρών θα πρέπει να ελέγξουν ε, μήπως ε, το εκτελεστικό τους ε, ε, λαϊλατεί αυτά τα χρήματα και τα κρύβει στις ε, ελβετικές τράπεζες. Μπορούν αυτά τα κοινοβούλια να ζητήσουν να ρωτήσουν τέτοιες σκληρές ερωτήσεις από τους υπουργούς που κάνουμε εμείς στη Δύση. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα κάναμε ένα μεγάλο καλό ώστε να μείνουν τα χρήματα αυτά σε αυτέ τι χώρε και να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη. Γιατί διαφορετικά είναι ένα φαύλο κύκλο. Εμεί βάζουμε τα λεφτά, μετά ξανάρχονται εδώ. Merci, cher Je donne la parole. Ε, ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφοι. Η κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Κρίστιαν Πρέντα που μας έδωσε μια τόσο καλή επισκόπηση των θεμάτων αυτών και τι θα βάλει στη γνωμοδότησή του. Ε, έχω και εγώ σημειώσει τα σημεία κριτικής που μας απασχόλησαν και προηγουμένως για τη Μεσημβρινή Αφρική και συμφωνώ απολύτως και χωρίς κανένα περιορισμό. Είπατε ότι θα πρέπει να δούμε τις χώρες αναπερίπτωση και να ε, παρατηρήσουμε τις, στις διάφορες ε, οικονομικές συμφωνίες στην εκάστοτε κατάσταση. Ε, έχετε το δίκιο και εδώ στην Ανατολική Αφρική τώρα πρόκειται για μια περιφέρεια που έχουμε τις τέσσερις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Από τις λιγότερο ανεπτυγμένες δηλαδή είναι τέσσερις. Βέβαια 25 χρόνια είναι μακρά χρονική περίοδος μεταβατική, αλλά 80% διάνοιξη της αγοράς για μια τέτοια χώρα μπορεί να είναι πάρα πολύ. Και ουσιαστικά, σύμφωνα με τους κανόνες ΠΟΕ, ΕΕ, οι χώρε αυτές που είναι λιγότερο αναπτυγμένες δεν θα πρέπει να ανοίξουν καθόλου τι αγροτικές του αγορέ. Εγώ σκέφτομαι τώρα λίγο την αγορά γάλακτος και κρέατος, δικιά μας, που σχεδόν έχουν καταρρεύσει, τι μέση είναι στο Ναδύρ και όλο λέμε να ανοίγουν καινούργιε αγορές. Ε, θυμάμαι πριν από 1,5 χρόνο, ένα χρόνο περίπου, στις Βρυξέλλες έκαναν μια εκδήλωση γαλακτοβιομήχανη και έκανε μια ομιλία ένας καθηγητής marketing, ο οποίος και τότε προφήτευσε ότι αν συνεχίσει να αυξάνεται σε εμά η γαλακτοπαραγωγή, που αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, κατά 6% οι ποσότητες δηλαδή, τότε θα πρέπει να δούμε πού θα εξάγουμε το γάλα μας και θα γίνει παιδική χαρά για τη γαλακτοβιομηχανία η Αφρική. Αυτό ακόμα το ακούω στα αυτιά μου ε, ως ε, παράθεση. Και αν ανοίξουν και άλλες αγορές, ε, ρωτώ με, την Αφρική σκεφτόμαστε όταν είναι τόσο μεγάλη πίεση για πού θα ε, ρίξουμε τα δικά μας πλεονάσματα Έχω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για αυτές τις ε, συμφωνίες εταιρικέ ε, σχέσεις. Ε, μήπως τις χρησιμοποιούμε και τις εκμεταλλευόμαστε για να εξάγουμε τις δικές μας υπερβολικές ποσότητες. Το ξέρω από την Κένια και την Βουρκίνα Φάσο αυτά στο παρελθόν και δεν θέλω να τα ξαναδώ μπροστά μου. Dann auch gesagt, dass wir einen starken Willen haben θέλετε, λέτε, να γίνει αυτή η συμφωνία μια καλή αναπτυξιακή συμφωνία. Μα εμείς στο Κοινοβούλιο δεν τα διαπραγματευόμαστε αυτά, ούτε μπορούμε να πούμε να βάλετε και το Α, να βάλετε και το Β. Ε, πολύ μεγάλη κριτική ακούγεται, αλλά δεν είμαστε σε θέση να το επιβάλλουμε, ούτε να το γράψουμε στη συμφωνία, ούτε να το διαπραγματευτούμε. Στο τέλο είτε ναι είτε όχι θα πούμε. Δηλαδή, προ όλη αυτή η συζήτηση. Εγώ έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση και αναγνώριση για όλη αυτή την κριτική, η οποία πέφτει, πάει στο βρόντο. Ούτε τον έλεγχο έχουμε αν θα επιβληθεί αυτό. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου πολύ μεγάλες για αυτή τη συμφωνία. Και πρέπει και εδώ να πω ότι η περιφερειακή ανάπτυξη στο εσωτερικό της Αφρικής θα πρέπει πρώτα να μεταξελιχθεί πριν αρχίσουμε να μιλάμε για αμοιβαία διάνοιξη των αγορών. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα σας παρακαλέσω να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Donc on attaque directement les questions. Ε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις σας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα ε, πρώτα απ' όλα για την ε, ευρύτατη περιγραφή αυτής της συμφωνίας. Προσβλέπουμε στη ολοκληρωμένη σας νομοδότηση. Ναι, ομοιομορφία είναι πολύ καλό σημείο, γιατί αυτό που ξεχνάμε είναι ότι ορισμένες από αυτές τις χώρες σύντομα θα είναι ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, στην κλίμακα του μέσου και ανώτερου εισοδήματος και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Ρουάντα και τη αργότερη Τανζανία. Αρχίζουν να σκέφτονται δεν θέλουμε να χάσουμε τα καθεστώτα duty free κτλ. Και οι ΕΠΑ θεωρούν ότι είναι ο τρόπος για να προχωρήσουν. Όμως η ομοιομορφία σημαίνει πως αυτές οι χώρες έχουν την πρόθεση να παρουσιαστούν στον κόσμο και όχι μόνο προς την Ευρώπη ως μπλοκ. Άρα λοιπόν δεν έχουμε επιλογή, θα πρέπει όλες να είναι σε μια συμφωνία. Το ίδιο είναι για την Κίνα, το ίδιο είναι και για τις ΗΠΑ. Είναι ενωμένοι, θέλουν να είναι σταθεροί, θέλουν να, να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι χώρες έχουν δημιουργήσει θεσμούς πολύ παρόμοιους με αυτούς της Ένωσης έχουν φανταστική ε, κοινοβουλευτική συνέλευση. Με όλο το σεβασμό για όλους σας ίσως και κάποιος ε, ακτιβισμός θα μπορούσε να αναζωογονήσει εκείνες τις ε, ε, κοινές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις που είχαμε με τους βουλευτές της Ανατολικής Αφρικής. Γιατί δεν γίνονται πια αυτά, αλλά εσείς σίγουρα μπορείτε να αναζωογονήσετε αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά λοιπόν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτή την περιφέρεια. Έχουν πολύ ισχυρά, ε, ισχυρά κοινοβούλια, είναι σημαντικό τα κοινοβούλια να έχουν φωνή και εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε αυτές οι κυβερνήσεις να περάσουν από, τη, ε, από τα κοινοβούλια. Το 2016 ήταν η ημερομηνία που προτάθηκε από το Κοινοβούλιο τότε, οπότε αυτή η ημερομηνία λέει υπογραφή και κύρωση, γιατί δεν είμαστε πια στο 2008 που δεχόμαστε μια, ε, μια κυβέρνηση που πάρει να παρακάμπτει το Κοινοβούλιο και να υπογράφει. Ε, ε αυτή τη φορά είπαμε θα πρέπει να περάσει από την κοινοβούλια σας. Ε, διαφορετικά δεν θα έχουμε συμφωνία. Ίσως να είναι πιο χρονοβόρο, αλλά εγώ είμαι βεβαία ότι θα είναι εκεί. Και έπειτα, απελευθέρωση. Απελευθέρωση θα είναι οι, οι, οι, οι μικρότερες δυνατές προσπάθειες που θα κάνουν. Μόνο το 16% σε 20 χρόνια, συν 2% σε 25 χρόνια. Ίσως το 2031 να είναι τελευταία ημερομηνία για το 80%, αλλά η συμφωνία θα συμφαρμοστεί πλήρως μόνο το 2041. Είναι το τελευταίο 2% αλλά έχει σημασία. Δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν. Είναι 25 χρόνια. Μιλάμε για περίπου το 60%. κάτω του πολλαπλασιασμού σα Είναι λιγότερο από 1% το χρόνο. Η ασυμμετρία λοιπόν υπήρχε. Σωστά την ανέφερε ο κύριος Πρέντα. Αλλά να τονίσω και πάλι ότι για, αυτόν την περιοχή, για αυτή την περιοχή οι κανόνες προέλευσης είναι πολύ, πολύ σημαντικοί και ο Βάνος, ο συνάδελφος που κάθεται δίπλα μου, ε, κοιτούσε ακριβώς ε, γιατί είναι πολύ σημαντικό τι κανόνες ισχύουν για αυτούς και τι κανόνες ισχύουν για μας. Υπάρχουν προϊόντα όπως και το ελαιόλαδο ας πούμε. Δεν το παράγουν αλλά ήθελαν να έχουν ε, το κανόνα και για το ελαιόλαδο αλλά και για τον καφέ. Οπότε βασικά πάμε πίσω στις αποκλεισμούς. Το γάλα αποκλείεται και όχι μόνο αποκλείεται αλλά αν μπει στους κανόνες μια δύνατον να εξαχθεί προς τις ε, χώρες αυτές με τις προτιμησιακές, ε, τα προτιμησιακά καθεστώτα. Δεν έχουν απελευθερώσει, αλλά έχουν πάει και για πολύ, ε, πολύ αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την προέλευση. Έπειτα, το θέμα του πώς φτάνουμε σε καλή παρακολούθηση του τμήματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θέλαμε να νερώσουμε τη συμφωνία του Κοτώνου που είναι υπέροχη και Θέλουμε να έχουμε μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να μπορούν να προστατευτούν και να ενεργοποιήσουν κυρώσεις. Οι ΕΠΑ έχουν, περιέχουν κυρώσεις, ενώ άλλες ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης όχι. Αυτό που είναι σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι εάν το κοτονού πέσει, εκπνεύσει, οι αρχές παραμένουν. Αυτό που παραμένει είναι η διαδικασία που περιλαμβάνεται στο Κοτονού υπό το άρθρο 96, σύμφωνα με την το οποίο πρέπει να μπει σε διάλογο κτλ. Και, και μάλιστα οι χώρε και πολλοί θέλουν να διατηρήσουν το Κοτονού, την συμφωνία του Κοτονού, γιατί έτσι δεν μπορεί μονομερός η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους ε, ε επιβάλλει τις κυρώσει που μπορεί να το κάνει αργότερα με τη βάση τη συνθήκη της Λισαβόνα άρθρο 145 και αυτό είναι η βάση για να επιβάλλουμε εμεί κυρώσει και να κλείσω δίνοντα σας τροφή για σκέψη το 97 είναι ένα άρθρο με τέλειε ε, διατάξεις περί διαφθοράς τέλειες. Είναι δικό μου σφάλμα που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Με μια έννοια έχουμε καλά μέσα που σήμερα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τα εκυβευόμενα θέματα από την ομοφοβία μέχρι την διαφθορά, την παιδική εργασία, αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Έκλεισε λοιπόν από δικιά μου πλευρά να πούμε ότι οι Αφρικανοί, Αφρικανοί αδερφοί μα έδωσαν όλα τα εργαλεία που θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μα για να προστατεύσουμε τι ευρωπαϊκέ αξίε, να προστατεύσουμε τα πιο σημαντικά από αυτά που θέλουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν και εμεί αξιόπιστα να ανταποκριθούμε σε αυτό και να πάω στην κατάσταση του Μπουρούντι. Έχουμε την ίδια κατάσταση, είχαμε την ίδια κατάσταση με τη Ζιμπάμπουε πριν από πολλά χρόνια, όταν εγώ ανέλαβα και είδα ότι για τη Ζιμπάμπουε δεν είχαμε στήριξη από τον προπολογισμό, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά, μπορούσαμε μόνο να στηρίξουμε τις ΜΚΟ σε αυτή τη χώρα. Άρα, κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Μπουρούντι. Τώρα μπαίνουμε στον διάλογο, με το άρθρο 8 Ο συνάδελφος που είναι ΔΕΦΚΟ είναι πολύ πιο εκτεθειμένος σε τέτοια πράγματα. Δεν στηρίζουμε πλέον ούτε τις αρχές του Μπουρούντι ούτε τίποτα με κανένα τρόπο. Ίσως να θέλει κάτι να προσθέσει. κύριος Δίβα εκτός μικροφώνου. Ε, πριν απαντήσει ο συνάδελφός σα γι' αυτό, αναφερθήκατε στο άρθρο 97. Τι πρέπει να κάνουμε για να ενεργοποιηθεί ή τι, να κάνουμε δηλαδή και ποιο πρέπει να κάνει κάτι για να λειτουργήσει. Υπάρχει διάταξη στη Συμφωνία Κοτονού και συμφωνώ με τη συνάδελφο Σάντρα ότι η διαφθορά είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και στην Αφρική και αλλού. Είναι πραγματικά πρόβλημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, στην ατζέντα της Αντίσα Μπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, όπου η διαφθορά ήταν ένα από τα θέματα τα βασικά που ε, είναι προβληματικά και αν θέλουμε να το συνδέσουμε με τις συμφωνίες ΣΟΕΣ θα χάσουμε τη σημασία του, συστήμα, ζητήματος μάλλον, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο σωστό πλαίσιο. Έγινε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για το πόσα χρήματα θα διατεθούν για την υποστήριξη της εφαρμογής ε, της ΣΟΕΣ και Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Βεβαίως έχουν απολύτως δεσμευτεί να το συνοδεύουν αυτό οικονομικά Εργαζόμαστε στα πλαίσια των διαδικασιών και των συστημάτων και βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για επιπλέον χρηματοδότηση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εάν δεν υπάρχουν ε, μεταρρυθμίσεις οικονομικές, δημοσιονομικές, ρυθμιστικές, πέντε χώρες. Δεν θα ε, τα λύσει τα προβλήματα η χρηματοοικονομική βοήθεια. Τι κάναμε λοιπόν, αξιολογήσαμε την κατάσταση με βάση τον ορισμό του ΣΑΓΙΑ, το Aid for Trade είδαμε όλα τα εθνικά εντεκτικά προγράμματα στο πλαίσιο του 10ου ΕΤΑ 1,4 δισεκατομμύρια εκτιμάται το ποσό που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο του 11 ΕΤΑ για τις πέντε χώρες αυτές για Aid for Trade, σύμφωνα με τον ορισμό DACTE του ΟΣΑ. Επίσης, από τα περιφερειακό ενδεικτικό πράγμα που έχουμε, ενδικό κενό και Δυτική και Ανατολική Αφρική 500 εκατομμύρια περίπου θα χρησιμοποιηθούν για αυτές τις πέντε χώρες που συζητούμε τώρα. Βέβαια μας ανησυχεί και μας ενδιαφέρει το να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση αυτών των ποσών, των σημαντικών ποσών. Γι' αυτό λοιπόν μόλις λάβαμε ε, μια συλλογική πρωτοβουλία, η ΔΕΛΤΑ ΤΡΕΙΝΤ, ε, η ΕΙΕΔ και η ΓΔ ΝΤΕΦΚΟ και ζητήσαμε τις πέντε αντιπροσωπείες μας ε, να ξεκινήσουν ε, να, εξετάζουν το δεχόμενο ενός ε, νέου κόνσεπτ σχέδια υλοποίησης ΣΟΕΣ για να μπορέσουν να ε, υποφεληθούν ε, των συμφωνιών αυτών από οικονομική πλευρά. Ε, και βέβαια με τα χαρά να επανέλθουμε εδώ για να σα δώσουμε περισσότερε λεπτομέρειε για αυτά τα σχέδια υλοποίηση ΟΕΣ. Δεν είναι μόνο για το πώ θα χρησιμοποιείται με το βέλτιστο τρόπο η οικονομική βοήθεια. Ο στόχο είναι επίση να υπάρχει ένα πραγματικό διάλογο για την οικονομική διπλωματία, πολιτικό διάλογο, επικοινωνίε, πληροφόρηση κτλ. Και Συνεργαζόμαστε με την Καμαλίτα Εμπόριο και η ΕΔ, άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Και επειδή είπατε να είμαστε σύντομοι, θα σταματήσω εδώ. Κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω κάτι, ότι ε, δεν ήθελα να μην απαντήσω, ε, να αλλά εμείς θέλουμε να υπάρχει μια συμμετοχική διαδικασία. Υπάρχουν ε, οι, όλες οι διαδικασίες και οι κυρώσεις, αλλά Μπορεί να μην χρησιμοποιήθηκαν εν μέρη τουλάχιστον καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι εμείς αυτό που συνεχώς ε, αναζητούμε είναι να έχουμε μία ε, δέσμευση και από αυτές τις χώρες ε, συμμετοχή τους. Φυσικά και κάθε συμφωνία οικονομικής τερκής πρέπει να αναλύεται με βάση τα υπέρ και τα κατά της ξεχωριστά. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη όμως ότι από πλευράς προσπάθειας λίγα κάνει αυτή η περιοχή για τις ΟΕΣ, γιατι δεν εχουν δέχουν μεγάλη απελευθέρωση, 65-66% ήδη είναι στο ε, στο μηδέν ε, για την Ινδία, για την Κίνα, για όλους. Άρα μας κάνουν πάρα μια ε, πολύ μικρή προσπάθεια, για μας μάλλον καμιά πολύ μικρή προσπάθεια που δεν είναι και τίποτα για αυτούς. Πρέπει να σας πω επίσης ότι θέλουν πραγματικά να έχουν μια συμβατική και όχι πλέον μονομερή ε, συμφωνία μαζί μας. Θέλουν δηλαδή να υπάρχει σύμβαση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα σταματήσουμε εδώ, θα ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτηση αφού ακούσουμε τον εισηγητή. Κύριο Πρέντα, επειδή πιέζει ο χρόνο, ε, να πω πολύ απλά ευχαριστώ όλου του συναδέλφου ε, και του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι παρεμβάσει του. Σε λίγο, σε λίγες μέρες, θα σα στείλω το κείμενο. Και θα κρίνετε από εκεί και πέρα με βάση την παρουσίαση, αλλά σίγουρα όπως ε, είπατε και εσείς δεν υπάρχουν τροπολογίες, ναι ή όχι πρέπει να πούμε, επειδή σε κάποιους συναδέλφους αρέσει να καταθέτω τροπολογίες, ε, βλέπω ότι λυπούνται, αλλά τι να κάνουμε. σε ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Επομένως, θα μας καταθέσει το σχέδιο γνωμοδότησής του ο εισηγητής στην συνεδρία μας στις 11 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο σημείο της σημερινής ημερησιάς διάταξης, εντολή για τον τριμερή διάλογο σε σχέση με το σχέδιο προπολογισμού 2017. ετήσιος προπολογισμό 2017 είναι το θέμα. Έχω μεγάλη χαρά που μπορώ να υποδέχομαι τον Γενικό Εισηγητή για τους προπολογισμού του 2017, τον συνάδελφό μας ε, Γένς Γκάιερ από την Επιτροπή Προπολογισμών. Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ένωσης ε, στοιχεί σε ένα σημαντικό ε, κομμάτι προπολογισμού, άρα είναι πολύ σημαντικό το έργο μας Εξού και είμαι πεπισμένος πως ο συνάδελφός μας Γιένς Γκάιερ θα ακούσουμε πολύ μεγάλη προσοχή της απόψης επιτροπής μας σε σχέση με τη, τα δημοσιογραφικά κονδύλια που αφορούν τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια. Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ μην μιλάμε να συνομιλείτε μέσα στην αίθουσα συντάκτη τη γνωμοδότηση ε, εκ μέρου τη Επιτροπή Ανάπτυξη, τον αδελφό μα Νίρι Ντέβα. Και του δίνω το λόγο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευτυχής που είναι εδώ ο εισηγητή ε, για τον προπολογισμό, ο κ. Γκάιρη. Είχαμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Θα του δώσω ένα πιο ενημερωμένο και πλήρε έγγραφο. Αλλά θα ήθελα να συμμεριστώ με την Επιτροπή κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε για τον προπολογισμό. Είναι σαφέ ε, μετά από την έκθεση του Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ότι το, τα χρήματα που υπάρχουν για τη διεθνή ανάπτυξη θα αυξηθούν 10 με 12 φορές παραπάνω από ό,τι ήταν πριν. Στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο είχαμε γύρω στα 15 με 16 δις να δαπανίσουμε στην Κομισιόν και άλλα 16 στο EDF στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ε, τώρα όλα μαζί ήμασταν ε, περίπου στα 14,8 με 16,8. Ε, δις. Εμείς όμως θέλουμε 300 δις να επενδυθούν μαζί με τους ιδιωτικούς εμερητές. και αυτά για να επενδυθούν όπου, εκεί όπου η, στην Αφρική και αλλού όπου η φτώχεια είναι ενδυμική και έχουμε γίνει εταίρες να αυξήσουμε τους όγκους εμπορίου και τις μεταποίηση και τις υπηρεσίες και ούτω καθεξής. οι ασφαλιστικές οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι υγειονομικές υπηρεσίες παρέχουν υπηρεσίες. Αν λοιπόν επενδύσουμε τέτοιου είδους χρήματα στην ενέργεια, την πράσινη ενέργεια, τις υποδομές, τις τηλεπικοινωνίες, τη γεωργία, το νερό, την ε, ε, παιδεία, την υγειονομική περίθευση, τα δικαιώματα, τα πνευματικά κτλ. κτλ θα δούμε τεράστια διαφορά στον κόσμο όπως ε, είναι σήμερα σε 5-10 χρόνια. Το συζητάμε τώρα εδώ και πολύ καιρό γιατί δεν μπορούμε να ζητούμε από τον Ευρωπαίο Φορολογόμενο να, τα, να πληρώνει ξανά και μανά. Όμω αν είχαμε το νέο ή αυτό τρόπο χρηματοδότηση, θα είχαμε εκατοντάδε δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πάνε στην ανάπτυξη και θα ήταν ένα ε, αθώος κύκλο γιατί πρόκειται για επενδύσει. και κάποια από αυτά τα χρήματα θα επανέλθουν. Και αν δημιουργηθεί ένα ταμείο ένα καταπίστευμα που θα μπορούν τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν εκεί. Σε 10-15 χρόνια δεν χρειάζεται να ζητάμε τίποτα από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Θα είναι ένας ε, ενάρετος κύκλος όπου χρήματα θα επενδύονται και θα αποδίδουν. Και ε, θα συνεχίζεται αυτή η αγαστή πορεία. The Commission is also working on a prospective EU-Africa investment plan which could be implemented through uh, public-private partnerships and θα είχαμε ωραίες ε, συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ΣΔΙΤ, και όλα θα πήγαιναν καλά. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε αυτό το τομέα είναι να δούμε πώς αυτός ο προπολογισμό για τούτη τη φορά, τούτη την περίοδο, θα μπορούσε να είναι διαφορετικός από ό,τι μέχρι τώρα. Να μπορέσουμε να αντλήσουμε και να οθήσουμε αυτές τις νέες δραστηριότητες. Πράγμα που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε έναν ιστορικό προϋπολογισμό, να πω στον συνάδελφο Γκάιερ, γιατί για πρώτη φορά θα βλέπαμε ένα διαφορετικό είδος Marshall Plan, ενό σχεδίου Marshall, που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά να είναι ένα είδος σχεδίου Marshall για την Αφρική, ένα επενδυτικό σχέδιο. Και ξέρω ότι τώρα πάω σε ολεστηρό έδαφος και ορισμένοι συνάδελφοι περιμένουν πώς και πώς για αλλά αν μπορούσαμε κάποια από αυτά τα χρήματα που μπαίνουν στο επενδυτικό σχέδιο να επιστρέψουν προς την Ευρώπη, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να συνεχίσουν να λειτουργούν τα εργοστάσια μας, δηλαδή να λειτουργήσει και προς όφελός μας, θα ήταν αμοιβαία σε αυτό το σχέδιο. Επενδύουμε Τα εργοστάσια μας δουλεύουν στο φουλ, πέφτει και ενέργεια και κερδίζουμε όλοι. και εδώ είναι το ληστηρό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι όταν δώσουμε, κάνουμε τέτοιες επενδύσεις σημαίνει ότι θα πρέπει να το δίνουμε με την προϋπόθεση ότι κάπως επανέρχεται σε μας. Οι Ιάπωνες το κάνουν αυτό εδώ και χρόνια. Δηλαδή όλες οι επενδύσεις τους ξαναποφέρουν. Και οι Κινέζοι το ίδιο κάνουν. Είμαστε οι μοναδικοί άνθρωποι στον κόσμο που δίνουν λεφτά και μετά φεύγουν αυτά για αλλού. Η απόδοση πάει στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στην Ινδία. Φτιάχτηκε ένα εργοστάσιο ποδηλάτων στην Ουγγάντα, το στήσαμε εμείς και οι πήραν τα κέρδη. Είμαστε τόσο large, τόσο κουβαρδάδες. Αλλά δεν λειτουργεί πια αυτό το σύστημα. Ε, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα βάλουμε ναι, λεφτά, αλλά θα κερδίσουμε και εμείς το κατητής μας. Πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε ώστε να μείνουν τα εστιατόρια... Τα... εργοστάσια μας να λειτουργήσουν και να αποφέρουν. In sustainable goals of the UN and I know that Christina Georgieva... Ήταν, ξέρω ότι η κυρία Γεωργίδα είπε στην, διάσκεψη, στην ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφή ότι πρέπει να καλύψουμε τα κενά χρηματοδότηση του κόσμου, αλλά σίγουρα αυτά που έχουμε εμεί στη διάθεσή μας δεν αρκούν. Έχουμε εκατομμύρια πρόσφυγες στη Συρία και γύρω, στις γύρω χώρες, στην Τουρκία, την Μέση Ανατολή. Τους βοηθάμε, αλλά κάποια φάση πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να τους επιστρέψουμε και αυτό θα χρειαστεί χρήματα. Και δεν ξέρουμε καν αν έχουμε τα χρήματα για να το καταφέρουμε αυτό. Αν θα βρούμε αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να επαναγκαταστήσουμε όλους αυτούς τους Σύριους πρόσφυγες και να προειδοποιήσω τους συναδέλφους ότι αν το ίδιο συμβεί που συμβαίνει στη Συρία συμβεί και στην Αίγυπτο, τότε ζήτω που καήκαμε θα πρέπει να μπορέσουμε να περιορίσουμε το ίσις και να σταματήσουμε την επέκτασή του και την προέλασή του. Τώρα, Τώρα, για άλλα θέματα για τον προπολογισμό, δεν έχω κάποια λεπτομέρειε να, πω, να συζητήσω με τον συνάδελφο, αλλά εν γέννη να πω ότι έχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις τρίτες χώρες. Έχουμε αυτές τις γραμμές του προπολογισμού. Σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με τον συνάδελφο και φίλο για τον προπολογισμό και ελπίζω ότι μέχρι ότου είναι η στιγμή να εγκριθεί, θα έχουμε καταφέρει να τα σκεφτούμε όλα αυτά, όλες αυτές τις νέες σκέψεις αυτή τη νέα πνοή, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι τελείω νέο. Merci, Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι, Ντεβα. Θα δώσω το λόγο τώρα στο συνάδελφο Ιένς Γκάιερ από την Επιτροπή Προπολογισμών. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το Νέρτζ Ντέβα για την ενδιαφέρουσα εισαγωγή. Σας θαυμάζω για τα οράματά σας, αλλά ακόμα δεσμευόμαστε από το δημοσιονομικό κανονισμό και τα σχέδια προϋπολογισμού που μας καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι να δούμε ε, τέλη του μηνός το σχέδιο προεπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορούμε να αξιολογήσουμε πόσα ε, έχουν ληφθεί υπόψη από τα όσα ενδιαφέροντα λέτε και φαντάζεστε. Γιατί η ειδική για την αναπτυξιακή πολιτική είναι εδώ, στη δική σας Επιτροπή, για να δούμε πόσα από αυτά που θέλετε μπορούν να μπουν στον προπολογισμό και να βρουν την πλειοψηφία της Επιτροπής σας. Προσωπικά, για τις ΔΙΤ έχω λιγότερα προβλήματα από ότι κάποιοι άλλοι για τα δημόσια οικονομικά που μπαίνουν σε ΔΙΤ. Αλλά κυρίω εγώ ασχολούμαι με τον προπολογισμό και ακόμα περισσότερο με τον έλεγχο του προπολογισμού. Και στις δύο λοιπόν αυτές ιδιότητες βλέπουμε συχνά ότι αυτό το μέσο αν μη τι άλλο χρειάζεται κάποια τελειοποίηση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ε, στις ε, προϋποθέσεις και στις φιλοδοξίες. Μπορεί να υπάρχουν ε, κάποιες σκέψεις για σημεία που λειτουργεί αυτό καλά, αλλά στον προϋπολογισμό του 2015 σίγουρα θα έχουμε και άλλα πάρα πολλά που εμπίπτουν στις δικές σας αρμοδιότητες και ενδιαφέροντα που μπορούμε Δεν θα μπορούμε να τα βάλουμε ακόμα στη ΔΙΤ. Από το 17 σίγουρα όχι. Αυτό το λέω έτσι. Αγαπητοί συνάδελφοι, πού βρισκόμαστε τώρα στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε ήδη το δεύτερο προγραμματικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ήταν ένα φυσιολογικό έτος, οικονομικό δηλαδή, σε σχέση με τα δημοσιονομικά και τη διαδικασία, κανονικά στην επόμενη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο θα έπρεπε να ψηφίσουμε την εντολή για το τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο για τα θέματα του προπολογισμού. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε σε μια τόσο κανονική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προπολογισμό, το σχέδιο της για το 2017 δεν το κατέθεσε στις 25 Μαΐου όπως είχε προβλεφθεί, αλλά βρήκε μια δικαιολογία εκεί πέρα ότι χρειάζεται ακόμα χρόνο για τον επαναυπολογισμό του κόστους για την προσφυγική κρίση και το ανέβαλε αυτό κατά ένα μήνα περίπου. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Η ανεπίσημη είναι ότι πρέπει να περάσει 23 Ιουνίου. Άρα το Βρετανικό δημοψήφισμα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύω. Η κασία είναι. Στον Περλεμόν φοβούνται να χτυπήσουν καμιά πόρτα, μήπως τρομάξει κανένας Βρετανός. Δηλαδή δεν κουνάνε τίποτα. Αλλά αυτά όλα μάλλον είναι, είναι φαντασία και έχει πραγματικότητα, ούτε πρόκειται να επεκταθώ σε αυτό. Αυτό δεν δημιουργεί αυτό κανένα πρόβλημα για μας, ουσιαστικό το, το Συμβούλιο θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει δεύτερο προγραμματικό έγγραφο, θα κάνουμε τα ίδια που κάναμε και το 2014, που ήμασταν εμείς τότε οι ε, ταραξίες γιατί είχαμε ευρωεκλογέ και είχαμε φύγει για τον προεκλογικό αγώνα μας και διακόψαμε 6 εβδομάδες τη δουλειά μας. Την ίδια διαδικασία θα υιοθετήσουμε λοιπόν με το 2014, που σημαίνει το εξής αν συμφωνήσουν και οι εκλεκτοί συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Προπολογισμών, θα στείλουμε μια συστατική επιστολή, recommendation letter, και οι γνωμοδοτήσει των επιμέρου επιτροπών θα συνηθούν έτσι ώστε οι Κομισιόν και το Συμβούλιο να έχουν μια εικόνα για το τι ε, πιστεύει και φρονεί το Κοινοβούλιο για τον προπολογισμό. Κατά τα άλλα, έχουμε ένα πρώτο προγραμματικό έγγραφο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον Απρίλιο το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε την πρότασή μου για τις ε, κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επ' αυτό να πω ακόμα μερικά λόγια, έτσι ώστε να έχετε μια εικόνα για το πώς εκτιμώ τη διαδικασία τη φετινή του προπολογισμού. Και πώς αποφάσισε το Κοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία. Κάτι που έχει σημασία και για τη δική σας Επιτροπή. Για τον προϋπολογισμό του 16, αυτόν που τώρα εκτελούμε, αλλά και για τον προϋπολογισμό του 15, τα μέσα για την καταπολέμηση της προσφυγικής κρίσης αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια και πλέον, για δύο χρόνια. Και σε αυτή την αύξηση ξεκάθαρα βλέπουμε ξεπεράσαμε τα όσα ζητούσε η Επιτροπή σας, ΔΕΒΕ. Δηλαδή κινητοποίησαμε σαφώς περισσότερα κονδύλια για την καταπολέμηση της προσφυγικής κρίσης και την υπέρβαση από ό,τι είχε ζητήσει και η δική σας Επιτροπή στη διαδικασία για τον προπολογισμό. Αυτά είναι στην κατηγορία 3, εσωτερική πολιτική και ε, Ευρώπη των πολιτών, όπου όλα τα μέσα είναι εκεί που έχουν να κάνουν με το άσυλο και ε, το Ταμείο το Σχετικό Ασύλου και Μετανάστευσης και είναι εσωτερική πολιτική της Ένωσης, αλλά και με την κατηγορία 4 που δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω γιατί τη γνωρίζετε εξαιρετικώς πώς. Αυτές τις αυξήσεις τις ζητούσε και η Επιτροπή και εμείς και ήμασταν απέναντι στο Συμβούλιο, το οποίο Συμβούλιο πάντα κινείται ανάμεσα στο ανώτατο όριο που μας βάζει το PDP το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το σημερινό επίπεδο του ευρωπαϊκού προπολογισμού θέλουν να έχουν όσο γίνεται περισσότερο περιθώριο λιγμών για πρόοπτα. Και εγώ ισχυρίζομαι ότι το κάνουν για να προστατεύουν τα εθνικά τους ταμεία, γιατί κυρίως πάντα οι καθαροί συνεισφορείς βγάζουν αυτό το επιχείρημα στις διαπραγματεύσεις. Όλοι οι υπόλοιποι τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βασανίζονται από αυτό το πρόβλημα και μάλλον θα ξαναδούμε αυτό το έργο. Τουλάχιστον έτσι διαβάζουμε το πρώτο προγραμματικό έγγραφο του Συμβουλίου. Όταν το πήρα, νόμιζα ότι καλά λάθος κάνανε και μου δώσανε τις guidelines του 15. γιατί στις τέσσερις πρώτες σελίδες μία, μία φράση είναι διαφορετική και μόνο στις δύο τελευταίες ε, σελίδες βλέπεις ότι είναι καινούριο το έγγραφο. Δηλαδή, στην σημερινή διαδικασία προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό που εκτελούμε τώρα έχουμε εξαντλήσει το ανώτατο όριο του PDP. Κανένα περιθώριο, μηδέν, τίποτα, δεν υπάρχει σάλιο. Και ρωτάω, εδώ μέσα υπάρχει κανένας που να μπορεί να επιχειρηματολογεί σοβαρά ότι θα έχει αλλάξει τόσο η κατάσταση το 17 ώστε να μπορούμε να έχουμε περιθώριο. Εγώ δεν μπορώ να το διαδώ αυτό και να πω ότι εντάξει Μπορεί κάποιο να μα πει ότι σε λίγου μήνε θα επέλθει και χειρία και κατάπαυση στο πυρό στη Συρία και θα γυρίσουν πίσω οι πρόσφυγε. Ψυχή. Άρα η σοβαρή πολιτική του προπολογισμού ε, προβλέπει συνέχιση της δύσκολης κατάστασης. Το Συμβούλιο τι κάνει, σου λέει αυτά που είπε και πέρσι, ότι τα περικόπτουμε αυτά, τα διαγράφουμε για να έχουμε περιθώριο για τις απρόοπτες δαπάνες. Νομίζω αυτό αγγίζουν την, τα όρια της μη ε, αντίληψης της πραγματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση πάρα πολύ ε, ενθουσιώδη και προσιλωμένη και η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών ταυτίζεται στις απόψει για την εκτίμηση κατάσταση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ θα τσακωθούμε με το Συμβούλιο και χοντρά και θα πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό και ε, ποντάρω πάρα πολύ στην υποστήριξη της δικής σας Επιτροπής, διότι οι κρίσεις συνεχίζονται και η οικονομική κατά τα άλλα δεν έχει ξεπεραστεί. Και θα κλείσουμε αυτό τον προπολογισμό σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να βρούμε πάνω από 4 δισεκατομμύρια από κάπου φέτος και του χρόνου έτσι ώστε να καλύψουμε την εγγύηση που συνδέεται με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ. Ναι, δηλαδή κάπου πρέπει να βρούμε τα δισεκατομμύρια για να αυξηθεί η εγγύηση για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ΕΦΣΙ. Και λέω το εξή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε κάνει συζήτηση στο Στρασβούργο όπου πολλοί συνάδελφοι ε, του Κοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ επικριτική. Γιατί η προσθετικότητα που είχαν τάξει δεν βλέπουμε να έρχεται. Και όλο και περισσότερο μας δημιουργείται η εντύπωση ότι με το νέο μέσο που με βρίσκει σύμφωνο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάνει αυτό που θα έκανε έτσι κι αλλιώς με την προσθετικότητα. Και σε σχέση με αυτό θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε πολύ προσεκτικά και είμαι απόλυτα πρόθυμος να το σκεφτούμε αυτό με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Προπολογισμών, τα χρήματα που έχουμε το κονδύλι για το ΕΦΣΥ να το βάλουμε στο αποθεματικό μέχρι να πληρωθούν ορισμένοι ε, όροι και προϋποθέσεις, δηλαδή να υπάρχει η προσθετικότητα, δηλαδή δεδομένη και να εξασφαλίζεται. Σε σχέση με αυτό, δεν θέλω να σας αποκρύψω το εξή. γιατί δηλαδή πρέπει να το πω. Κύριε Ντέβα, τα κράτη-μέλη και το δικό σας και το δικό μου ε, χάρηκαν πάρα πολύ για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο ε, που δεν ε, αυξήθηκε, για πρώτη φορά αλλά μειώθηκε. Και μάλιστα συνέχεραν ο ένας τον άλλον ε, που έχουμε λιγότερα χρήματα από ό,τι στο παρελθόν για τους στόχους μας και μας παρηγόρησαν λέγοντας ότι έχουμε τώρα χρηματοδοτικά μέσα που θα κάνουν μόχλευση και δεν συμμαζεύεται. Αλλά αυτό ισχύει, ε, εδώ ισχύει αυτό που είπα στην αρχή ότι δεν μας πείθουν πάρα πολύ. Συμφωνώ επί της ουσίας, αλλά δεν με έχει πείσει αυτό. Συμφωνώ θεωρητικά. Πάντως τα λεφτά είναι λιγότερα. Τώρα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και την αναγνωρίζουμε όπου οι κρίσεις σοβούν γύρω-γύρω και αυξάνονται και οξύνονται και τα κράτη-μέλη δεν κατεβάζουν καμιά καλύτερη ιδέα από το να λένε ότι αν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κρίσει, θα επιτεθούμε πρώτα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όσο και να είναι. Γιατί τώρα θα το πω ε, ηρωνικά και ε, με κάποια κακία. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κολυμπάει στα λεφτά και δεύτερον δεν ξέρει τι να τα κάνει. Αυτά λένε στις πρωτεύουσες. Αυτά ε, είναι πραγματικά ε, λάθος. Ε, ε, κινδυνεύει να εκραγεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν προκύπτει από κάπου ένα κενό, μια τρύπα, πάμε και τα παίρνουμε από αλλού για να τη βουλώσουμε και δημιουργούμε μια άλλη. Από το 2013 έχουμε τις κρίσεις και δεν περιμένουν και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, που διαπραγματευτήκαμε ήταν για τον καλό καιρό. Ε, μπορεί για το 2013 να ήταν καλό που ήταν ε, το κλίμα εύκρατο και ηλιόλουστο, αλλά για το 2016 και για το 2017 δεν υπάρχει. Ποτέ δεν βρέθηκε τέτοιος προπολογισμό που να μπορεί να λειτουργεί όπως το έχουν σκεφτεί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Δεν είναι όμως πρόθυμοι στο τέλος του τους να ελέγξουν, να αναθεωρήσουν το PDP, αλλά συνεχίζουμε τα γνωστά. Και έχω την αίσθηση ότι δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Και αυτή είναι η πρόταση επίσης, ε, πρόταση του Κοινοβουλίου από τις κατευθυντήριες γραμμές, να αυξήσουμε τα κονδύλια που έχουμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να το συνδέσουμε με τις οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια οικονομική ε, προσέγγιση και πρόβλεψη. Το 2015 έκανε ας πούμε την έκθεση για την ανάπτυξη. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο, μην νομίζετε ότι συμφωνώ 100% ως πολιτικές προθέσεις ένα προς ένα. Αν το κάναμε αυτό, θα μας παρέλειε και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Οικονομική Αρχή. Απλώς να αναλύσουμε, να δούμε τι μπορούμε να υιοθετήσουμε, τι μπορούμε να ζητήσουμε από άλλα θεσμικά όργανα, να προσανατολίζεται κάπως ο, ο εκεί ε, για να αυξηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό με χαρά να το κάνω. Και επίση έχουμε και κάποιες άλλες προτάσεις. Τα κέντρα βάρους από τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 βλέπε καταπολέμηση της ανεργίας που με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί είμαι και σοσιαλδημοκράτης, ιδιαίτερα η ενεργεία των νέων. Είχαμε την πρωτοβουλία για την εργασία των νέων. Θα πρέπει να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική βεβαίως, αλλά δεν γίνεται χωρίς επιπλέον λεφτά αυτό. Βάζεις πολιτικούς στόχους, πρέπει να βάλεις και το χέρι στην τσέπη για την καταπολέμηση της φτώχειας. Για ένα τελευταίο ε, που θέλω να το βάλω και στον προπολογισμό για να κλείσει εδώ ο κύκλος ε, προς εσάς κύριε αυτό που είπατε στην αρχή. Η Επιτροπή προβληματίζεται για κάτι το οποίο λέγεται performance-based budgeting, δηλαδή προϋπολογισμός βάση επιδόσεων, είπε πραγμένο. Έχει δίκιο. Εγώ ε, κάνω έλεγχο προϋπολογισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αν το συνδέσουν με το Ταμείο περιφερειακή Ανάπτυξης, α πούμε, φτιάχνει το Ταμείο περιφερειακή Ανάπτυξης μια γέφυρα. Τα πάντα ήταν άψογα, ο διαγωνισμός, η προκήρυξη, το κόστος, οι προθεσμίε στηρίθηκαν τα πάντα, Ωραία, ε, στη συμμόρφωση αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά αν η γέφυρα είναι φτιαγμένη σε λάθο μέρος και δεν τη χρησιμοποιεί κανεί, τότε δεν είναι η επίδοση καλή. Άρα θα πρέπει να προβληματιστούμε όχι μόνο πω θα βελτιώσουμε τις διαδικασίες και τη συμμόρφωση, αλλά εάν πιάνει τόπο το έργο και αν χρησιμοποιείται και πώς ε, βελτιώνουμε τι επιδόσει. Αυτό συζητούμε τώρα. Δηλαδή, μπορεί καταρχήν το έργο που προτείνει ο Ντέβα ή το μέσο να είναι το σωστό, αλλά μπορεί και όχι. Και ένα τελευταίο, και θα κλείσω εδώ. Η Επιτροπή σας Να το πω αλλιώς. Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορείτε, τι μπορείτε να μας προτείνετε για να έχουμε επιτυχία στο Συμβούλιο των Υπουργών Αναπτυξιακής Βοήθειας και πώς μπορούμε να τα μετρήσουμε αυτά συγκεκριμένα για να έχουμε και επιχειρήματα για τη βοήθεια, για την ανάπτυξη αλλά και για την καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ευχαριστώ πολύ. Σας κύριε Γκάιερ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιότητες εισηγητές. Καταρχάς στον κύριο Λίτς. Ναι, ναι. Κύριε Χαουταλά. Ζητώ συγγνώμη κυρία Χάουταλα, χρειάστηκε να πάει σε επόμενη συνάντηση που έχει να πάρω το λόγο, αν θέλετε, αν συμφωνείτε, ξενόματός της. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Τώρα είναι δύσκολο κανείς να συζητήσει για κάτι που δεν έχει στα χέρια του. Και όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταθέσει σχέδιο προπολογισμού, τι να το κάνουμε. Είναι λίγο τώρα χαρτορίχτρα η ιστορία αυτή. Πάντως αυτό που είπατε είναι πολύ σπουδαίο, ότι αυξήθηκαν τα κονδύλια για την προσφυγική κρίση και το μεταναστευτικό. Αν κατάλαβα καλά, μιλήσατε για 10 δις για τη διετία 15-16. Και εδώ έχω μια μεγάλη ανησυχία. Θα έχουμε μεταφορά πόρων από ε, τα δημόσια αγαθά, τα παγκόσμια ή από το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Από εκεί θα τα πάρουν και από εκεί ανησυχούμε κι εμείς. Είναι λίγο παράδοξο αυτό. Γιατί κάναμε τη συμφωνία αυτή των Παρισίων μόλις και χρειαζόμαστε τα κονδύλια στις χώρες για να εφαρμοστεί. Και άμα μιλάμε για μετανάστευση και προσφυγιά, η κλιματική αλλαγή χρειάζεται καταπολέμηση γιατί είναι μία από τις αιτίε. Για να μπορεί ο κόσμος να παραμένει στον τόπο του και να έχει μέλλον και προοπτική και κάποια ελπίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε από εκεί χρήματα. Και αν κάνουμε οικονομίες για να χρηματοδοτήσουμε κάτι ε, ε, έκτακτο στην Ευρώπη, δεν είναι σωστό. Παρακαλώ αυτό να σας προβληματίσει και να το φροντίσετε. Και ένα δεύτερο, να έχετε υπόψη σας, στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι το θέμα των προϋποθέσεων και των συνθηκών που επικρατούν στα στους καταβλισμούς προσφυγικούς. Ήρθε μια τεράστια προσφυγική ροή. Η κατάσταση ε, επιδεινώθηκε μαζικά. Δεν είχαν σχολεία για τα παιδιά τους στους καταβλισμούς εκεί και χάνονται ολόκληρες γενιές. Μεγαλώνουν τα παιδιά χωρίς να έχουν καμία ελπίδα για το μέλλον τους. Παρακαλώ να το προσέξετε και να κοιτάξετε και τι κονδύλια χρειάζονται από ποιες θέσεις του προπολογισμού. Είναι αφόρητες και απαράδεκτες οποιασδήποτε περικοπές εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Σάιφος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τώρα κυριαρχεί το θέμα, αριθμών ένα αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Στην ενδιάμεση αναθεώρηση θα πρέπει να δούμε ποια είναι ε, τα θέματα αυτά και πώς θα προσαρμόσουμε τις ανάγκες στην πραγματικότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να προσπαθούμε να βοηθούμε επιτόπου. Εγώ πήγα στον Καζιαντέπ στην Τουρκία και στους προσφυγικούς καταβλισμούς μου είπαν οι άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν σπίτια τους. Για ποιο λόγο στον Καζιαντέπ κάθε πρόσφυγας παίρνει μια πιστοτική ε, κάρτα που τους βάζουν 30 ευρώ το μήνα, είναι τα δύο τρίτα των όσων χρειάζονται για να επιβιώσουν. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και επιτόπου για να μπορεί ο καθένας να ζει 100% όχι κατά δύο τρίτα. Η τουρκική κυβέρνηση λέει ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε ο κόσμος να βγαίνει από τους καταβλισμούς και να ε, δουλεύει και πηγαίνουν και στις εταιρείες και στα ε, κτήματα για να δουλεύουν και να βγάλουν και το κάτι Αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε και εκείνους που στην Τουρκία ε, προσφέρουν ε, μαθήματα. Μάλιστα μαθήματα γλωσσών κάνουν σε αρβικά, τουρκικά, ευρωπαϊκές γλώσσες. Θα πρέπει η Επιτροπή Ανάπτυξης να επενδύσει ε, στις διαπροσωπικές ε, σχέσεις, μικρή εταιρεία προς μικρή εταιρεία. Όσο πιο μικρές είναι οι δομές που συνεργάζονται, τόσο καλύτερα λειτουργούν ε, οι εταιρικέ σχέσεις. Οπότε θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε ποια είναι εκείνα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε. Τον Έρασμο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Έχουμε τόσα πολλά προγράμματα ισχυρά που χρησιμοποιούμε οι ίδιοι για να αυξήσουμε ε, ε, τις δυνατότητές μας και να καλύψουμε τις διαφορές με στρατηγικό τρόπο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η δική μας Επιτροπή Ανάπτυξης ε, μαζί με την Επιτροπή Προπολογισμών να ψάξουν νέες προτεραιότητες και να βοηθηθούν γι' αυτό. Κατά των διακινητών δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέπεται Ε, όσο αλλάζουμε την πολιτική μας, ε, τόσο περισσότερα λεφτά βγάζουν διακινητές. Θα πρέπει να αυξήσουμε ε, τις νόμιμες οδούς, με διαφάνεια και νομιμότητα να έρχονται οι άνθρωποι στην Ευρώπη, να έχουν σωστή στέγαση, σωστή εργασία για να μπορούν να ζουν και αξιοπρεπώς. Και η διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνεται νόμιμα και το αίτημα για νέε στρατηγικέ και για νέου στόχου είναι θεμητό. Και αν δεν το, αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιο θα το κάνει αυτό στη θέση μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρασαλόμ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω το Γέννη πρώτα απ' όλα. Γέννη, ε, μας ε, έκανες ε, ένα μάθημα για τον προϋπολογισμό. Ένα εξαιρετικό μάθημα. Και όχι μόνο αυτό, Βέβαια, μας έδωσες και μία όχι τόσο αισιόδοξη εικόνα για το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της Ένωσης από πλευράς προϋπολογισμού. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ μόνο στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πράγματι, οι συνάδελφοί μου που μίλησαν πριν από εμένα ήδη τόνισαν την ανάγκη να διαθέσουμε επαρκείς σπόρους για την ανθρωπιστική βοήθεια και θα ήθελα να τονίσω κάτι που και εσύ Γέννης ανέφερες, ότι δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει έλλειψη προβλεψιμότητας σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο για πρόβλεπτα Ακριβώς διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα απαιτεί προβλεψιμότητα, άρα ασφαλεί σίγουρους πόρους. λίγου πολλού πάντως σίγουρους. Επομένω, ε, η παράγραφος 4, μάλλον η κατηγορία 4 του προπολογισμού θα πρέπει να είναι επαρκώ ε, περιφοκοδοτημένη. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, θέλω να πω ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα πρέπει να τίθεται υπό όρους. Οι αρχές της ανθρωπιστικής δράσης λένε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η παροχή βοήθειας ε, στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη να υπόκειται σε πολιτικές προποθέσει και όρους. Εντάξει, αλλά ε, σε άλλες περιπτώσεις ναι, όχι ανθρωπιστική βοήθεια όμως. Ανθρωπιστική, μάλλον αναπτυξιακή βοήθεια τώρα. Τα ταμεία, τα, τα αναπτυξιακά κονδύλια δεν θα πρέπει να καλύπτουν ανάγκες που άμεσα ε, δεν αφορούν την ανάπτυξη. Ή έχουν να κάνουν με την κρίση της φτώχειας. Δηλαδή δεν θα πρέπει η αναπτυξιακή βοήθεια επίσης να συνεισφέρει στην έλεγχο των συνόρων. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ανήκει αλλού. Δεν θα πρέπει να υπάρξει αυτή η παράκαμψη. Δηλαδή να βγάζουμε κονδύλια από, αυτό το, από αυτή τη γραμμή του υπολογισμού με την ασφάλεια του συνόρων κτλ. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά το δύσκολο του εγχειρήματο. Πρέπει να διαπραγματευτεί με την Κομισιόν, με το Συμβούλιο και να διαπραγματευτεί επίση με όλε τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ εδώ. Κάθε μία θα σου λέει ότι η δική του στόχη είναι η προτεραιότητα, η απόλυτη προτεραιότητα κλιματική αλλαγή, διεθνές εμπόριο, γεωργία, αλληλεία και ούτω καθεξής. Όμως, για ένα είμαι βέβαιος. Και φαντάζομαι ότι και η δική σου πρόταση και επιθυμία είναι ήτι να εφαρμόσουμε τις αξίες μας στην πράξη απέναντι σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση που ζει τόσος πολλοί κόσμος εντός και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Το λόγο τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γάμα δέλτα ντεύκο, γάμα δέλτα έκο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι. Μίλησε συνάδελφος πριν για μάντις ε, και κρυστάλλινες σφαίρες. Πράγματι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τις χαρτορίχτρες ούτε τους ε, μάντις. Διότι υπάρχουν οι λόγοι που ε, είπε ο κύριος Γκάγερ, γνωστή ή μη γνωστή, είναι αυτή που έκανα να μην έχει γίνει ακόμη δεκτό το σχέδιο προπολογισμού και να μην έχουμε και την πρόταση της Κομισιόν πριν τα τέλη του μήνα. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια βασική γραμμή, είμαστε στη φάση προγραμματισμού. Ο προπολογισμός λοιπόν που θα κατατεθεί ε, θα ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με το PVP και τον προγραμματισμό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Πράγματι, το είπατε όλοι νομίζω, είμαστε αντιμέτωποι με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, από τη μια πλευρά, να αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση, αλλά και από την άλλη πλευρά, να συνεχίσουμε να ε, υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε αυτά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Νομίζω το είπαν όλοι οι βουλευτές. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε τα χρήματα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη για άλλους σκοπούς, για βραχυπρόθεσμες δράσεις, για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης τώρα. Βέβαια, σίγουρα τα χρήματα που προορίζονται για την ανάπτυξη είναι για μακροπρόθεσμους ε, σκοπούς, γιατί αλλιώς η κρίση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο και θα έχουμε όλο και περισσότερους πρόσφυγες στο μέλλον. Άρα, έξω και ζητήσαμε και πρόσθετα κονδύλια. Θα την τελευταία ανακοίνωση για τη μετανάστευση, εξωτερική πτυχή. Εκεί αναφέρουμε κάποια ποσά τα οποία θα θέλαμε να μας διατεθούν για να συνεχίσουμε τις δράσεις που έχουμε αναλάβει. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, για να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα Ε, την κρίση και να φέρουμε σε πέρα τις δράσεις που έχουμε να φέρουμε σε πέρα. Έχουμε τον DCI, τον Μέσο Αναπτυξικής Συνεργασίας, χώρες σημαντικές όπως Πακιστάν, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές καλύπτονται από το μέσο αυτό. Σίγουρα όλοι έχουμε το μυαλό μας και στη Σύρια και τους πρόσφυγες που οι μετανάστες από την Αφρική ή τη Σύρια. Όμως, να μην ξεχνάμε και το Αφγανιστάν, που είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες ε, που σοβούν κρίσει. Είναι σημαντικό λοιπόν και το έργο που κάνει ο συγητής. Μπορεί να μην υπάρχει απλή οδοξία ελπίδα όμως υπάρχει. Να Απευθύνουμε στον κύριο Ντέβα τώρα. Πράγματι, εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στο, στην διευκόλυνση επενδύσεων για τη Λατινική Αμερική, για την Ασία, την Αφρική. Έχουμε σχετικούς μηχανισμούς, άρα μπορούμε ε, να πούμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί για επενδύσεις και λειτουργούν, λειτουργούν καλά. Και υπάρχουν και εις ε, που λειτουργούν επίσης καλά. Όλα όσα είπατε, σίγουρα δεν λέω ότι είναι η υπάρχουν όμως και τα επεξεργαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Εδώ ολοκληρώνω εγώ και δίνω το λόγο στο συνάδελφο από τη ΓΔ Αντεύκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που έχω να πω είναι πολύ σύντομο, θα είναι πολύ σύντομο γιατί υπόθηκαν τα πιο πολλά. Θα είναι πάνω στην ανθρωπιστική βοήθεια σίγουρα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου το μέγεθος, η διάσταση της κρίσης είναι τεράστια και υπερβαίνει κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους. Δεν θέλω να προκαταλάβω το σχέδιο προπολογισμού που θα καταθέσει τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι από ό,τι αναμένουμε, τουλάχιστον ε, στις αρχές ε, του έτους δεν θα έχουμε τα ίδια ποσά στον προπολογισμό όπως για το 2016. Και το 2015 και το 2016 υπήρχαν πακέτα για να αντιμετωπίσουμε τις ε, την προσφυγική κρίση 200 εκατομμύρια το 2015 και άλλα 300 το 2016. Και αυτό τα ποσά τη δυνατότητα στην Κομισιόν και ε, τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία να αντιμετωπίσει άλλε κρίσει, όχι την προσφυγική, άλλε κρίσει, χωρίς να επηρεάσει η τρέχουσα προσφυγική κρίση, τις άλλες. Σίγουρα είχαμε μια πολύ μεγάλη κρίση που όμως δεν είχε δραματικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αντιμετώπιση άλλων κρίσεων στον κόσμο. Όπως είπαν σήμερα οι βουλευτές, και στον προπασμό και στην ενδιάμεση αξιολόγηση που θα γίνει, δεν θα έχουμε μάλλον αυξήσεις θα έχουμε μια επανεξέταση όμως των προτεραιοτήτων και από ό,τι φαίνεται θα δοθεί έμφαση ιδίω σε ζητήματα όπως είναι απλούστευση, μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερα παραδοτέα αποτελέσματα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, μείωση διοικητικών δαπανών για παράδειγμα, βέλτιστη δυνατή χρηματοοικονομική βοήθεια προς τους ε, τελικούς δικούς κτλ. Αυτά είχα να πω και συμφωνώ απόλυτα με ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Γκάιερ. Έλα, θα σας παρακαλούσα να μην μιλήσετε πάνω από πέντε λεπτά, γιατί ήδη είμαστε σχεδόν εκτός χρόνου. Πέντε λεπτά παρακαλώ και άλλα πέντε στο συνάδελφο Ευχαριστώ. Σύνολο δέκα. Έχετε το λόγο κύριε Γκάιε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ το πεντάλεπτο νομίζω. Συμφωνώ επί της ουσίας στα σημαντικότερα θέματα που είπαν οι συνάδελφοι και με τη συνάδελφο Χόιμποχ. συμφωνώ ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα από τον προπολογισμό ε, να μειωθεί το ε, DCI για να πάνε αλλού τα λεφτά για την καταπολέμηση της προσφυγικής κρίσης. Σας είπα ότι για να βουλώσουμε τρύπες κόβουμε αλλού το ύφασμα ε, ε, έχουμε μια καινούρια τρύπα για μετά πάμε να μπαλώσουμε κάτι άλλο ε, και δημιουργείται πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ανώτατο όριο στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο επέβαλε ειδικά μέσα που εμείς λέγαμε over and above, δηλαδή πάνω από την οροφή, είναι επιπλέον κονδύλια. Το Συμβούλιο το ερμηνεύει διαφορετικά. Ε, αν συνεχίσει λοιπόν να το ερμηνεύει έτσι, δεν θα έχουμε καινούριο φρέσκο χρήμα και θα πρέπει να είμαστε ευφυείς στις ε, μεταφορές πιστώσεων ε, από τη μια κατηγορία στην άλλη. Τώρα, οι ανθρωπιστικές συνθήκες στους καταβλισμούς, τον έφερε και ο Ερίκε και η κυρία Χόιμπουχ, αυτό είναι εκ των όνων κάνευ όρος για την καταπολέμηση της κρίσης, ε, της προσφυγικής. Εκεί θα πρέπει να βοηθήσουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε και θα ε, είναι και ο μεγαλύτερος μοχλός για τη βοήθεια. Ερίκε, ζήτησες ανθρωπιστική βοήθεια επαρκή εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε στο βαθμό που προχωρούμε. Ε, θα αγωνιστούμε να υπάρχουν αρκετά κονδύλια στην ανθρωπιστική βοήθεια και η θέση του Κοινοβουλίου αυτή θα είναι, θα, θα θέλησουμε να εξαντλήσουμε το ανώτατο όριο της κατηγορίας 4 για να πάει ένα μεγάλο κλάσμα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Τελευταία πρόταση, διότι έχει σημασία σε σχέση με αυτό και πιστεύω ότι είναι της δικής σας επιτροπής, τουλάχιστον προς ενημέρωση να το πω εδώ. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ από τη στάση των κρατών μελών για τα καταπιστεύματα. Δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο στο δημοσιονομικό κανονισμό έτσι ώστε για να βρούμε χρήματα από τον κοινοτικό προπολογισμό, από ε, τον προπολογισμό των κρατών μελών, από τη δική τους αναπτυξιακή βοήθεια για να τα συνανθρήσουμε και να έχουμε μοχλό. Τι βλέπουμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της, δίνει τα κονδύλια για το καταπίστευμα και για τη διευκόλυνση για την Τουρκία ισχύει το ίδιο, με διαφορετικό τρόπο λένε το ίδιο μέσο και τι βλέπουμε, τα κράτη-μέλη ε, κάνουν το χαζό. Όχι όλα, πολλά κράτη-μέλη βοηθάνε πάρα πολύ, τουλάχιστον Γερμανία και ε, Βρετανία ξέρω ότι διμερώς κάνουν πολλά. Απαιτούν να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μέσο, αλλά δεν το χρησιμοποιούν μετά οι ίδιοι. Και εγώ δεν πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει τους λογαριασμούς που κάνουν τα κράτη-μέλη. Ε, εάν δεν είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο τα κράτη-μέλη, τότε για ποιο λόγο να δεσμεύσω κονδύλια περισσότερο σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από εκείνα που προτίθεται και διατίθεται τα κράτη να δώσουν. Εάν τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν αλλάξουν την τακτική τους για τα καταπιστεύματα, τότε στο μέλλον θα Επελευθερώνω τόσα κονδύλια όσα απελευθερώνουν τα κράτη-μέλη. Ένα προς ένα. Εάν και 28 μαζί βάζουν 50 εκατομμύρια στο καταπίστευμα, άλλα τόσα θα είναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όχι εμείς θα κάνουμε ότι υποσχεθήκαμε 250, όχι. Θα βάλουμε και εμείς 50 να δούμε τι θα γίνει. Και αν φύγουν αυτά τα 100, δαπανηθούν, θα πρέπει να συζητήσουμε για τη μελλοντική μας τάση. Ε, συμφωνώ με αυτό το μέσο των καταπιστευμάτων, αλλά με μεγάλη δυσφορία και με αυξημένη και αυξανόμενη πικρία. Βλέπω τα κράτη-μέλη να κάνουν διάφορες εξαγγελίες και μεγαλώστομε στη Βαλέτα, στην Άγκυρα ε, και όταν έχει ώρα να βάλουν το χέρι στη τσέπη ε, τα λουριά και τα, και τα και αυτό με εκνευρίζει. Και είναι και ανεύθυνο το να περίπτει ο ένας ευθύνη στον άλλον. Και θα πρέπει να καταλάβουν κάποια στιγμή και τα Υπουργεία Οικονομικών ότι δεν είμαστε εδώ το μακρύ χέρι των κρατών μελών ή ο πάγκος εργασίας, η επέκτασή του, ότι είμαστε κάτι άλλο και θα πρέπει να το καταλάβουν. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Το λόγο για κύριο Δέβα. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν συναρπαστική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων σε όλου του συναντέλφου μου και ιδίω βέβαια στον κύριο Γκάιερ αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να ευχαριστήσω για τις απόψεις της σε σχέση με τις διάφορες πτυχές. Συμφωνώ απολύτω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει να υποκλέπεται. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη και να γίνεται ανθρωπιστική βοήθεια, διότι δεν έχουμε χρήματα για ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί έτσι τι κάνουμε, επιδεινώνουμε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα και θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερα μεταναστευτικά ρεύματα ή ρεύματα προσφύγων γιατί οι χώρε του δεν μπορούν να του κρατήσουν αυτού του ανθρώπου, δεν μπορούν να του εξασφαλίσουν απασχόληση, ούτε καν τα προστοζή. Πρόκειται για έναν παύλο, φαύλο κύκλο που θα μπορούσαμε να τον κάνουμε έναν ενάρετο κύκλο. extraordinary in trying to Ο κύριος ε, Γκάιερ κάνει ό,τι μπορεί για να ε, βγάλει από τη μύγα ξύγκη. Τώρα, λυπούμε, αλλά πρέπει να σας θέσω ένα ερώτημα και σας δω και τον προτέρων συγγνώμη. Αλλά ξέρετε, έμεινα ύπνος δύο-τρεις μέρες, επειδή με ανησυχεί πάρα πολύ το τι θα γίνει την Πέμπτη. Υπάρχει ένας ελέφαντας ε, στο δωμάτιο. Κάνουμε ότι δεν τον βλέπουμε. Υπάρχει όμως ελέφαντας αυτός στο δωμάτιο και μπορεί να τα κάνει όλα λίμπα αν δεν αλλάξει τίποτα τις επόμενες λίγες ημέρες. Και δεν ξέρω προς τα που οδεύουμε με αυτό το καταραμένο το δημοψήφισμα. Αλλά τέλος πάντων Υπάρχει αυτό το δημοψήφισμα. Ερωτώ λοιπόν, έχετε προπολογισμό σε περίπτωση ανάγκης, γιατί θα βρεθείτε με 18 δι ε, παραπάνω, γιατί είναι λίρε 20 δις τρύπα, αν δεν πάει καλά το πράγμα. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των παιδιών που βρίσκονται στου καταβλισμού, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Ή θα δημιουργήσουμε άλλη μια γενιά προσφύγων που δεν θα μπορούν κάπου να εγκατασταθούν και να δουν δουλειά, ή θα κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι ουσιαστικά Είμαστε όλοι ε, ε, στο ίδιο μήκο κύματο, ε, αλλά είναι δύσκολη καιρή και δεν είναι εύκολο να σχεδιάσουμε αυτόν τον υπολογισμό. Και για αυτό καταλαβαίνω γιατί δεν έχει υποβάλει ακόμη σχέδιο προπολογισμού η Κομισιόν, ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είμαστε και από του καθαρού εισφορεί άλλωστε εμεί. Η Βρετανία εννοώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεβά. Η απάντηση θα δοθεί διμερός φαντάζομαι από το Γιάννης Γκάιερ διότι είμαστε εκτός χρόνου. Λοιπόν, ήθελα να σας πω μόνο ότι είναι το τελευταίο θέμα αυτό για απόψε. Αύριο ραντεβού εδώ θα έρθει ο Επίτροπος κύριος Στυλιανίδης για τη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης 22-23 Μαΐου. Αύριο το πρωί ραντεβού. Καλό σας βράδυ.